είναι ενημέρωση για την απόφαση των συντονιστών. Η κυρία Γκουλάρ από την Άλντε να γίνει συγγήτρια για την, επιτροπή, την έκθεση της ΕΚΟΝ για την αναθεώρηση ε, του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης ε, στο πλαίσιο ε, του ΣΥΚΣΠΑΚ και του ΤΟΥΠΑΚ. Συμφωνήσαμε με τον κύριο να μην μιλήσουμε για το άρθρο 54 Συνδεδεμένη Επιτροπή, αλλά να είμαστε το όργανο υποβολής της έκθεσης σαν να ήμασταν υπό το άρθρο 50. Επομένω, η κυρία Γκουλάχ θα προσκληθεί σε συνεδριάσεις των σχιωδών και θα ήθελα οι συνάδελφοι από την Άλντε να ελέγξουν κατά πόσο αυτό λειτουργεί καλά και για τις τροπολογίες συμφωνήσαμε και λάβαμε τη δέσμευση ότι οι τροπολογίες που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της ΑΦΚΟ ε, θα διέπονται από το άρθρο 54. Δηλαδή θα υπάρχει ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ θα δούμε αν θα τηρήσουν αυτή τη δέσμευση. Όμως η κυρία Γκουλάχ είναι η συγγήτρια εκ μέρους μας. Να περάσω τώρα στο σημείο 5. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 7ης Ιουλίου. Βεβαίως ε, είναι στη διάθεσή σας και θεωρώ ότι έχουν εγκριθεί, εκτός και αν υπάρχει αντίσταση μάλλον κάποια αντίθετη γνώμη μέχρι το τέλος ε, της ε, συνεδρίασης. Σας ενημερώνω επίσης ότι ε, προβάλλεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση αυτή. Τώρα, περιμένουμε τον προσωρινό πρόεδρο του Συμβουλίου, κύριο Σάντρο για να μας ενημερώσει. Ah, Βρίσκεται ακόμα στην αίθουσα πρωτοκόλου. Χρειάζεται λοιπόν ακόμα μερικά λεπτά. Υπενθυμίζω ότι η Ιταλική Προεδρία αποφάσισε να διοργανώσει ομάδα υψηλού επίπεδου με εκπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο της ομάδας ε, φίλη της Προεδρίας κατά τη διάρκεια της τελικής Προεδρίας λοιπόν για να εργαστούν επί της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα. Και αυτή η απόφαση συζητήθηκε και, και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ε, του Αυγούστου, όπου μας εκπροσώπησε η κυρία Σπινέλη. Και το Σεπτέμβριο είχαμε και τη δική της ε, οπτική γωνία και γνώμη. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Γκόζη για να μας πει τι καινούργιο υπάρχει σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αρμοδιότητας της ΑΦΚΟ. Θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Επειδή ο κύριο Υπουργό Γκόζη θα πρέπει να φύγει στις 5 παραδέτου το αργότερο ή απλώ ε, διορθώστε με αν ε, τα λέω λάθο. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο, παρακαλώ αμέσως μετά την παρουσίαση να μας ε, το, να μας το πούν και θα δούμε πόσο χρόνο έχουμε. Ο Ρίτσαρ Κόρμπερ προφανώς μας έχει εξηγήσει. Κύριε ε, Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που δίνετε στην ε, Προεδρεύουσα χώρα και σε εμά, έτσι ώστε να συζητήσουμε για μία ακόμα φορά θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει, είχαμε μάλλον αναφέρει και στην ε, ε, αρχική μας συνάντηση εκεί είχαμε αναφέρει τις προθέσεις της Προεδρίας δηλαδή να ξεκινήσουμε μια συζήτηση όσον αφορά την λειτουργία των θεσμών και η συζήτηση αυτή ξεκίνησε ε, μάλιστα πρέπει να πω ότι ξεκίνησε και ένα πιο επιχειρησιακό κομμάτι ε, και γι' αυτό ακριβώς ήρθε εδώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω δηλαδή πρώτα πώς ε, προχώρησαν τα ζητήματα στην στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 17ης Αυγούστου. Εκεί είπαμε πώς θα ξεκινήσει το υπηρεσιακό κομμάτι και μάλιστα η Επιτροπή σας και εσείς ε, ε, κυρία Πρόεδρε εκπροσωπηθήκατε από την συνάδελφα κυρία Μπάρμπαρα Σπινέλη. Μετά θα ε, αναφερθώ στις ε, διεργασίες ε, της ομάδας φίλη της Προεδρίας, καθώς επίσης και την, τις αναφορές που έκανα στο τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Όσον αφορά τη συζήτηση την οποία ξεκινήσαμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, εκεί προέκυψαν ορισμένα θέματα. Ας πούμε, ε, κάποια διτά ζητήματα τα οποία, ή κάποιες αρχές ε, στις οποίες θέλησαν οι συνάδελφοι να εντάξουν τη δραστηριότητά μας. Η πρώτη στα πλαίσια της ε, Προεδρίας μας λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δεκέμβριο δηλαδή η Προεδρία θα πρέπει να υποβάλει ε, μία έκθεση στην, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Εκεί αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε τις ε, συζητήσεις μας στα πλαίσια των ε, ισχυουσών συμφωνιών και συνθήκων. Η μεγάλη πλειοψηφία των αντιπροσωπιών αποφάσισαν να μην ανοίξει το θέμα της ενδεχόμενης μεταρρύθμισης των συνθήκων. Επίσης, απεφασίστη να οργανωθούν οι εργασίες γύρω από τέσσερα θέματα τα οποία αφορούν και τέσσερις επιχειρησιακές συνεδριάσεις οι οποίες ε, ασχολούνται ακριβώς με αυτά τα τέσσερα θέματα. Πρώτον, ε, στην πρώτη συνεδρία ήταν αυτή η εισαγωγική ε, η οποία αφορούσε μια συζήτηση για το πώς λειτουργικά, επιχειρησιακά δηλαδή, οι εργασίες πολιτικού περιεχομένου μπορούν να ενσωματώσουν κάποια ευρωπαϊκά ζητήματα τα οποία ε, είχαν ε, ε, μεγάλο αντίκτυπο στην σε την νομοθετική εργασία. Αναφέρομαι στην επικουρικότητα εδώ και στην αναλογικότητα. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα οι σχέσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και οι ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και το, το κράτος. Τρίτο σημείο είναι αυτό το οποίο ονομάζεται governance, διακυβέρνηση, υπό το φως κάποιων ε, κυρίως προσφάτων ε, πολιτικών που αφορούν κυρίως ε, οικονομικά ζητήματα. Τέταρτο θέμα εστίασης θα είναι το πώς και πόσο χρησιμοποιήθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή με με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε το δυναμικό, όπως λέμε, της ε, συνθήκης της ε, Λισαβόνας στα πλαίσια των διαφόρων πολιτικών και επίσης πόσο ε, μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. η συζήτηση σε διπουργικό επίπεδο ε, ήγηρε για κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να θίξω εδώ ενώπιόν σας. Το πρώτο βεβαίως είναι και άλλωστε σας ευχαριστώ ε, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να είμαι εδώ. Ε, το πρώτο λοιπόν ήταν να αξιολογήσουμε τη διαθεσμική συμφωνία του 2003, Better Law Making. Το, η καλύτερη, το καλύτερα νομοθετή, πούμε. Επίσης, η αξιολόγηση μιας ε, ενδεχόμενης νέας διαπραγμάτευσης, νέας συζήτησης για, το, ε, για τη Συμφωνία Πλαίσιο του 2010 αφορά ε, και την δικιά σας Επιτροπή, γιατί πολλές αντιπροσωπείες θεώρησαν ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί μία ενδεχόμενη συμμετοχή του Συμβουλίου. Ένα άλλο σημείο αφορά εξέταση του πώς λειτουργούν οι τριμερείς διάλογοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σε γενικό επίπεδο απασχολεί τους πάντες, δηλαδή όσον αφορά την διαφάνεια της φάσης αυτής και όσον αφορά ε, γενικότερα την ευρωπαϊκή ε, διαδικασία νομοθέτησης. Ένα άλλο σημείο είναι ο ετήσιος και πολυετής νομοθετικός προγραμματισμός. Δηλαδή, εάν και κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια όσον αφορά ε, τον νομοθετικό προγραμματισμό, έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Τώρα θα ήταν η καταλληλότερη περίοδος ε, τώρα που ξεκινάει ένας νέος πολιτικός κύκλος, μια νέα πολιτική περίοδος. Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα καθώς επίσης και ο ρόλος του ε, Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων όσον αφορά την προετοιμασία ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η δυνατότητα ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα να προτείνονται στον Προεδρεύοντα ε, κάποιες προτάσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το θεματολόγιο, όσον αφορά την ατζέντα και επίσης, και επίσης η παρακολούθηση το follow-up ε, και η υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, αυτά είναι τα γενικά θέματα, τα κεντρικά θέματα τα οποία εφήγησαν από τις διάφορες αντιπροσωπίες. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, αποφάσισε μετά από προσπάθεια και προσπάθεια πυθούς μάλιστα, περισσότερο στις Βρυξεόλες και λιγότερο ε, ε, στις πρωτεύουσες, γιατί πρέπει να σας πω κυρία Πρόεδρε, ότι ε, λιγότερη αντίσταση βρήκαμε στις πρωτεύουσες για να ξεκινήσει ένας τέτοιος διάλογος και περισσότερο, περισσότερη αντίσταση διαπιστώσαμε στις Βρυξέλλες. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα θέμα ταμπού επομένως προηγουμένως από τις ε, πρωτεύουσες και νομίζω ότι είναι καλό να το λέμε ε, γιατί ίσως μερικές φορές ο δρόμος που ενώνει τα διάφορα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες είναι πιο δύσβατος εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, ε εν πάση περιπτώσει δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να το συζητήσουμε αυτό, απλώς ήθελα να το αναφέρω έτσι ακροθυγώς. Έλεγα λοιπόν ότι επιμείναμε και δημιουργήθηκε η ομάδα φίλων της ε, Προεδρίας επί τη βάση των εργασιών που έγιναν και στο παρελθόν και επομένως αυτή η ομάδα των φίλων ε, της ε, Προεδρίας η οποία αναφέρεται στην Κορεπέρ και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ήδη συνεδρίασε μία φορά και συζήτησε ακριβώς κάποιες γενικές αρχές, δηλαδή ε, πώς υλοποιούνται, πώς εφαρμόζονται ε, τα στοιχεία κλειδιά, αυτά τα οποία ε, συνδέονται με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα που ήδη ανέφερα προηγουμένως. Από αυτήν την άποψη όλες οι αντιπροσωπείες δεν θεώρησαν απαραίτητο να ξανατεθεί το ζήτημα τροποποίησης αυτών των αρχών, αλλά μόνο ε, το θέμα της ε, βελτίωσης. Θεωρούν λοιπόν ότι η υλοποίηση δεν θα πρέπει ε, διαρκώς να περιλαμβάνει λιγότερη ευρωπαϊκή δράση, αλλά να περιλαμβάνει καλύτερη ευρωπαϊκή δράση. Αναπτύχθηκε μια πρώτη συζήτηση λοιπόν γύρω από αυτήν την αρχή της επικουρικότητας και μερικές αντιπροσωπείες μάλιστα είπαν ότι καλό θα ήταν να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να αξιολογήσουμε στο εσωτερικό της, στα πλαίσια λοιπόν της ε, ε, νομοθετικής ε, προετοιμασίας και του νομοθετικού προγραμματισμού αυτήν την αρχή της επικουρικότητας και ενδεχομένως να δούμε το κατά πόσο θα ήταν καλό να έχουμε στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων μια ετήσια συζήτηση, μια συζήτηση σε ετήσια βάση. Ένα άλλο θέμα το οποίο ανεδίθη και το οποίο συνδέεται με τις ε, αξιολογήσεις αντικτύπου, αυτή δηλαδή την αξιολόγηση αντικτύπου που ακολουθεί τις νομοθετικές προτάσεις ε, ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί πολλές ήταν οι αντιπροσωπείες οι οποίες είπαν ότι ίσως καλό θα ήταν να μην γίνονται μονάχα αξιολογήσεις αντικτύπου στην αρχή όταν ξεκινάει η πρόταση από το Κολέγιο των Επιτροπών αλλά και αργότερα και με τους δύο συνομοθέτες γιατί μετά από τις τροποποιήσεις ε, που ε, ξεκινούν ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο πολλές φορές αλλάζει η αρχιτεκτονική και νομίζω ότι αυτή η αξιολόγηση ίσως θα μπορούσε να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό την υποβάλλω σαν ε, ε, ζήτημα σε εσάς. Ένα άλλο θέμα, ε, ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Επ' αυτού οι διάφορες αντιπροσωπείες φρονούν ότι το ισχύον πλαίσιο από θεσμικής και νομικής απόψεως είναι ικανοποιητικό, αλλά υπάρχουν και σημεία τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Δηλαδή η υλοποίηση είναι ελλειπής και θα πρέπει να ξεπεράσουμε την απλή νομική κοινωνική ας πούμε υλοποίηση και θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς την περισσότερο πολιτική υλοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ε, να κάνουμε και διάφορα πρακτικά ζητηματάκια, να λαμβάνουμε υπόψη μας το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου, ε, γιατί υπάρχουν άλλα κοινοβούλια τα οποία συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι συνεδριάζουν με διαφορετική ε, χρονική συχνότητα, άλλες φορές το Κοινοβούλιο είναι εδώ, άλλες φορές είναι σε ολομέλεια κτλ. Θα πρέπει όλα αυτά τα πρακτικά ζητήματα να ληφθούν υπόψη και ε, ε, υπάρχει αίτημα για μεγαλύτερη παρουσία των επιτρόπων στα εθνικά κοινοβούλια. Ένα άλλο θέμα το οποίο εφήγει είναι το θέμα των στόχων των συνθήκων. Ε, έγινε συζήτηση σχετικά με την δυνατότητα ή το σκόπιμο της κατάρτισης προτεραιοτήτων μεταξύ των στόχων των ε, ε, συνθήκων. Υπάρχουν κάποιες αντιπροσωπείες οι οποίες ε, λένε ότι θα πρέπει όλους τους στόχους να τους επιδιώκουμε για να τους υλοποιούμε τον ίδιο τρόπο. Άλλοι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ιεράρχηση, άλλοι ότι θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση αντικτύπου και ορισμένες αντιπροσωπείες θεωρούν ότι σε αυτή την πολιτική συγκαιρία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κυρίως τα άρθρα 8 και 9 ε, της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνουμε κυρίως υπόψη τον αντίκτυπο των νομοθετικών ευρωπαϊκών προτάσεων ε, σε θέματα όπως είναι η καταπολέμηση των ανισοτήτων, όπως είναι η ανεργία, η απασχόληση ε, όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Ε, ξέρουν ε, οι κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε αυτή την ιδιαίτερη πολιτική στιγμή. Τελευταίο σημείο και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία έθεσε και το ζήτημα της αρχής της αλληλεγγύης η αρχή της αλληλεγγύη ε, ε, στις συνθήκες αναφέρεται περίπου 20 φορές, ε, είτε για το άσυλο, είτε για τη μετανάστευση, είτε για οικονομικούς στόχους. Σε όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρεται και η αλληλεγγύη, η αρχή της αλληλεγγύη, και η οποία ε, σύμφωνα και με την αρχή και με τις ε, αρχές της Προεδρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να εντάσσεται περισσότερο στη στρατηγική και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε συζήτηση ε, για αλληλεγγύη όσον αφορά και την κλιματική αλληλεγγύη, το άσυλο, την μετανάστευση, κάποιες, κάποια ειδικά σκέλη της γεωπολιτικής ή της κοινή πολιτικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής ε, επίσης ε, ε, αναφέρθηκε το ότι αντίθετα από άλλες αρχές η αρχή της ελληνικής δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με οριζόντιο τρόπο αλλά αναπερίπτωση. Είναι δύο, διαφορετικές, είναι δύο διαφορετικά στοιχεία τα οποία η Προεδρία θεωρεί σημαντικά και τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να βάλει στην τράπεζα των συζητήσεων. Αυτά ε, συζητήθηκαν λοιπόν. Η επόμενη συνεδρίαση, η συνάντηση των φίλων της Προεδρίας θα λάβει χώρα τη 10η Οκτωβρίου και λεπτομερέστερα θα ε, ε, μελετήσει θέματα και αν βεβαίως εσείς το επιθυμείτε μετά μπορώ να έρθω να αναφερθώ σε εσά σχετικά με τα όσα θα έχουν συζητηθεί εκεί. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ ήταν ο πρώτος ο οποίος ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που παίρνω την πρώτη θέση, αλλά πρέπει να φύγω για να πάω σε μία από τις ακροάσεις όπου είμαι εισηγητής. Ζητώ συγγνώμη, λοιπόν, θα είμαι πολύ αγενής, θα σας ρωτήσω και μετά θα φύγω και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι οι φίλοι της Προεδρίας είναι βέβαια μια εσωτερική ομάδα του Συμβουλίου. Αλλά όπως ξέρετε από την εμπειρία σας, οι καλύτεροι φίλοι του Συμβουλίου είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι στους οποίους πρέπει να βασίζεστε και γι' αυτό είσαστε εδώ. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα εμποδίσει την ευκαιρία από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας προσφέρουμε τις δικές μας απόψεις και τα σχόλιά μας για τις πρωτοβουλίε που ξεκινάτε. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι χαίρομαι για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει αλλάξει γνώμη και αποφάσισε ότι πρέπει και αυτό να προσχωρήσει τη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπογραφεί εδώ και μερικά χρόνια μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου. Τουλάχιστον αυτή είναι η κίνηση του Συμβουλίου. Κάλλιο αργά παραποτέ θα σας έλεγα. Ίσως επιτέλους το Συμβούλιο αναγνωρίζει το ότι το Κοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν είχαν δίκιο να προσπαθήσουν να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους στις διαθεσμικές με ένα τέτοιο τρόπο και αν θέλετε να υπογράψετε, να προσυπογράψετε αυτό το κείμενο, ακόμα και να το βελτιώσετε, όχι βέβαια να το αποδυναμώσετε, αυτό θα είναι κάτι ιδιαίτερα καλόδεκτο για μα. Για τα σημεία που προτείνετε να εξετάσετε, θα σας πρότεινα να είσαστε λίγο πιο επιφυλακτικός. Καταρχήν, οι αρχές της απόδοσης, της επικορικότητος και της αναλογικότητας. Μπορεί κανείς να τα συνοψίσει όλα αυτά ως μια ανταπόκριση σε φόβους ότι γίνεται υπερσυγκεντρωτική ή υπερυθμισμένη η υπεριθυμισμενη η Ένωση. Όταν τώρα όμως οι εθνικές κυβερνήσεις εκφράζουν τέτοιου είδους ανησυχίες, μερικές φορές κάποιοι υπουργοί, ιδίως σε χώρες, μας δίνουν την εντύπωση ότι οι Βρυξέλλες μας επιβάλλουν πάρα πολύ γραφειοκρατία, κανόνες και οι ίδιοι υπουργοί δεν έχουν ιδέα για όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που ξυπνάνε και βλέπουν ότι οι Βρυξέλλες τους τα έχουν επιβάλει. Αλλά βέβαια δεν μπορεί να εγκριθεί κανένα νομοθέτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μονάχα με, χωρίς την έγκριση όχι μόνο αυτού του εκλεκτού κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου. Και ποιο είναι σε αυτό το Συμβούλιο αυτοί οι ίδιοι υπουργοί, αυτέ οι ίδιε εθνικέ κυβερνήσει, οι οποίε μετά γκρινιάζουν για την Κομισιόν. Είναι υπουργοί που είναι μέλη εθνικών κυβερνήσεων και υπόλογοι σε εθνικά κοινοβούλια. Και χρειάζεται και μια ευρεία πλειοψηφία. 74% των ψήφων στο τωρινό σύστημα στάθμισης χρειάζονται για να μπορέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει οποιοδήποτε νομοθέτημα με ενισχυμένη με ειδική πλειοψηφία. Τίποτα δεν περνάει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν δεν υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία των κρατών μελών που συμφωνεί ότι αυτό είναι απαραίτητο και συμφωνούν για το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσίας. Κάποια από αυτά τα παράπονα λοιπόν εγώ τα παίρνω με μια πρέζα αλάτι όπως λέμε στα αγγλικά. Βέβαια πολλές φορές οι ορισμένοι υπουργοί μπορεί να παρασύρονται από το ευρωπαϊκό πνεύμα τους γητεύει η Κομισιόν με την ευγλωτία της και δέχονται πράγματα τα οποία μετά μετανιώνουν. Δεν με πείθει τώρα το επιχείρημα αυτό για να είμαι ειλικρινής. Από τότε που εισαγάγαμε το, τη διαδικασία της, ε, ε της κίτρινης κάρτας και της Πορτοκαλή κάρτας για να μπορούν να παρεμβαίνουν τα εθνικά κοινοβούλια, ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε η πορτοκαλί κάρτα από τα εθνικά κοινοβούλια. Μόνο δύο περιπτώσεις υπήρξαν όπου υπήρξε επαρκή υποστήριξη για μια κίτρινη κάρτα και σε μια από τι δύο περιπτώσει, η Κομισιόν απέσυρε την πρότασή τη ούτω ή άλλω. Στη δεύτερη περίπτωση ήταν θέμα ενισχυμένη συνεργασία, οπότε εναπέκτω σε αυτούς οι οποίοι θέλανε να συνεργαστούν, να συνεργαστούν και δεν χρειάστηκε να αποσυρθεί μια πρόταση. Δύο περιπτώσει σε πέντε χρόνια. Αυτό δεν μου δείχνει μια ένωση η οποία πηγαίνει προς μια υπερσυγκεντρωτικότητα ή υπερβολική υπερβολικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και αν λέτε να βελτιωθεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων, ναι, αλλά όχι για την επικουρικότητα, για τυπικά θέματα, αλλά για θέματα ουσίας. Έχουν ένα διάστημα 8 αποφάσεων προτού το Συμβούλιο σταθμίσει τη θέση του να εξετάσουν τις νομοθετικές προτάσεις, προτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις εξετάσει, Αυτές οι 8 εβδομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα Εθνικά Κοινοβούλια, όχι μόνο για να ελέγχουν κατά πόσον υπήρξε σεβασμός της αρχής επικορικότητας, συνήθως γίνεται αυτό, αλλά να δούνε και την ουσία και να συζητήσουν με τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος θα του εκπροσωπεί στο Συμβουλίο Υπουργών, πρωτού πάει στην Βρυξέλλε, πρωτού έρθει στην συνάντηση των Υπουργών. Όχι να του τα ψέλουν εκ των υστέρων. Μερικά κοινοβουλία το κάνουν ήδη αυτό. Τα βαλτικά κράτη, οι σκανδιναβικέ χώρε είναι πρωτοπόροι σε αυτά. Κάποια άλλα κοινοβούλια θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν αλλαγέ των ευρωπαϊκών κανόνων και σίγουρα δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι συνθήκε. Μία τελευταία παρατήρηση. Αναφερθήκατε στους στόχους που βρίσκονται στο προήμιο. Στη χώρα μου υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι θα πρέπει να επαναξετάσουμε τους στόχους που αναφέρονται στο προήμιο των συνδικών για μια όλο και πιο στενή προσέγγιση, μια όλο και πιο στενή ένωση. Όλο το, το όλο και πιο στενά σημαίνει για αυτούς ότι θα στενεύει όλο και θα στενεύει αυτή η ένωση και στο τέλος θα έχει ζουληθεί σε ένα υλικό σημείο. Αυτά όμως δεν έχουν νόημα. Αν διαβάσετε αυτά που λέει μετά η συνθήκη, λέει ότι οι αποφάσεις βάσει αρχή αρχής της θα πρέπει να λαμβάνονται εκεί που είναι πιο κοντά στου πολίτε. Αυτό είναι πιο ισορροπημένη άποψη. Αν διαβάσετε λοιπόν το σύνολο, είναι έτσι. Βέβαια δεν διαβάζουν όλο το κείμενο πολλοί υπουργοί στη δική μου χώρα και γι' αυτό θέλουν να ξαναγράψουν τι συνθήκε, δηλαδή παντού ομοφωνία, παντού εθνική επικύρωση για να φύγει και αυτό το οποίο βρίσκεται στο πρόημο. Ούτως ή άλλως αυτή είναι μια δήλωση προθέσεων, τίποτα παραπάνω. Αλλά παρόλα αυτά θέλουν να το σβήσουν από τις συνθήκες. Ελπίζω ότι θα αντισταθείτε σε μια τέτοια τάση. Θα έχετε και παιδαγωγικό χαρακτήρα έναντι ορισμένων υπουργών που έρχονται στις ε, συναντήσεις σας και όχι να φύγουμε σε μια κατεύθυνση η οποία δεν ωφελεί κανένα. Ευχαριστώ. Ε, αν σε παρηγορεί δεν είναι μοναχα οι δικοί σου που λένε κάτι τέτοιο. Ο Τζο Σέφριν τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ. Με μεγάλη χαρά σας ξαναβλέπω εδώ. Και ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά και πλήρη αυτά που μας είπατε. Κάποιες τώρα σκέψεις ή ερωτήματα που πλησιάζουν αρκετά αυτά που είπε ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι το κεντρικό ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα, γιατί τουλάχιστον από εκεί που βρίσκομαι, βλέπω να υπάρχει μια μεγάλη απόκληση μεταξύ πολιτικών και οικονομικών πραγματικότητων στην Ευρώπη, που ελπίζω ότι και οι φίλοι της Προεδρίας συζητούν αυτό το πρόβλημα. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες συζητήσεις σε σχέση με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αλλά την Παρασκευή ήμουνα σε μία συνδιάσκεψη στην ε, Βουδαπέστη μεταξύ κοινοβουλευτικών της περιοχής του Δούναβη και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Και ίσως αυτά που τους έλεγα τους έδωσαν την εντύπωση ότι είμαι εξωγήινος. Δεν ξέρανε τι ήταν αυτά που λέγαμε, που έλεγα. Ενδεχομένως υπήρχε μία άγνοια από τη μεριά τους, ενδεχομένως μία συγκεκαλυμμένη εχθρότητα σε αυτά που είπα, αλλά αυτό το οποίο τους είπα ήταν αυτό που του, σας είπε προηγουμένως ο Ρίτσαρ Κόρμπετ. Να συναντιέστε με τους υπουργού σας πριν από ένα συμβούλιο και να ζητάτε πληροφόρηση και να τους δίνετε την άποψή τους. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τύχει περισσότερες Έμφαση και οι επίτροποι θα, θα πρέπει να έρχονται σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων για να ενημερώνουν τους βουλευτέ. Και πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό η δική μας επιτροπή, μάλλον συγγνώμη, η τρέχουσα επιτροπή είναι πιο ανοιχτή σε κάτι τέτοιο από την προηγούμενη επιτροπή, δηλαδή οι επίτροποι να πηγαίνουν και να εργάζονται και σε εθνικό επίπεδο και να συζητούν εκεί. Εάν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό το πράγμα, τότε γίνεται και πολιτικό θέμα και αρχίζει να πλησιάζει περισσότερο την κοινή γνώμη και τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Το πλαίσιο λοιπόν των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια μπορεί να είναι νομικά ικανοποιητικό, από πολιτική έποψη όμως είναι ελληματικό. Υπάρχουν χάσματα σε οποιαδήποτε διμερή σχέση, ακόμα και αν είναι ε, πολυμερείς αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες περαιτέρω εξετάσει και ιδέε, αλλά θα έπρεπε να κάνουμε πραγματικά αμοιβαία καλύτερη τη σχέση αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Κοινοβουλίων. Κάτι άλλο που δεν αναφέρατε, τουλάχιστον εγώ δεν το έπιασα, ήταν η πρωτοβουλία πολιτών, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δεν ξέρω αν είναι αυτό στη δική σα αρμοδιότητα, αλλά σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να είναι, ή τουλάχιστον οι φίλοι τη Προεδρία θα πρέπει να το εξετάσει. Εμεί είχαμε μακροσκελέστατε συζητήσει για το θέμα αυτό στο προηγούμενο Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί πολύ καλά αυτό το εργαλείο όμως. Μπορούμε να συζητήσουμε και να έχουμε διαφωνία για το γιατί δεν γίνεται, δεν λειτουργεί καλά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε γιατί έχει δυνατότητα να κινητοποιήσει μεγάλους αριθμούς πολιτών και να τους κάνει να συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη παρατήρηση στο θέμα της λογοδοσίας που είπατε. <clears throat> Πράγματι υπάρχουν κενά στο θέμα αυτό και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για το πώς πρέπει να τροποποιηθεί. Και το τελευταίο, πάλι έρχομαι στο θέμα της επικουρικότητας. Μόνο μια ιδέα σας δίνω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα διαρθωτικού χαρακτήρα. Περισσότερη επικουρικότητα σημαίνει περισσότερη πολυμορφία. Και αυτό μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη έλλειψη συνοχής. Και αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε και αυτό είναι μια δυσκολία που την αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Γιώ Λάινεν, αν είναι έτοιμο. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Είναι κάπως το σύνθημα της νέας θητείας η καλύτερη νομοθεσία. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν σημαίνει λιγότερη Ευρώπη, αλλά καλύτερη νομοθεσία αλλά έχουμε ένα πρόβλημα και στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο. Είπε ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ ότι χρειάζεται 74% των ψήφων για να υπάρχει μια ειδική πλειοψηφία και εμεί χρειαζόμαστε κάποιε πολιτικέ ομάδε, άμα θέλουμε να έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι μια επιτροπή που έχει πολύ νομοθετικό έργο και υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις πλειοψηφίες. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το εξετάσουμε, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε και το έργο της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος με το να υπάρχουν λιγότερες ε, ε, εκθέσεις οι οποίες υπερφορτώνουν αυτή την Επιτροπή ίσως λιγότερη νομοθεσία για το περιβάλλον, λιγότερη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και λιγότερη υπερλεπτομεριακή νομοθεσία. Χαίρομαι που είπατε ότι είναι εντάξει το νομικό πλαίσιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οι συνθήκες είναι πολύ σαφείς για τις αρμοδιότητες των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Και πράγματι δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα, υπάρχει η κίτρινη κάρτα και εν ανάγκη η πορτοκαλί. 1η Δεκεμβρίου θα γίνει στη Ρώμη η επόμενη συνεδρίαση της ΚΟΣΑΚ, όπου θα τεθεί το θέμα της υπερεθνικότητας και της δημοκρατίας. Θα είναι στην ημερησία διάταξη. Και εκεί κάποιοι θα αγωνιστούν για να έχουν και κόκκινη κάρτα και όχι μονάχα κίτρινη και πορτοκαλί ε, Αλλά εδώ πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε <clears throat> τη διαδικασία. Αντίθετα θα πρέπει να βελτιώσουμε στην πράξη τη διαδικασία που ακολουθείτε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κόκκινη κάρτα. Μια τρίτη παρατήρηση. Είπατε ότι υπάρχουν δυνατότητες, μάλλον ότι έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της συνθήκης της ε, ε, Λισαβόνας, εκτός από θέματα όπως αυτά που είναι η ενισχυμένη συνεργασία. Υπάρχουν ρήτρες αυτού του είδου, Αλλά μπορεί να έχει το Συμβούλιο μια πρόταση προς εμάς και να μας εξηγήσει ποιες είναι οι περαιτέρω διατάξεις της Συνδίκης Λισαβόνας που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην πράξη. Ευχαριστώ. Άλλος ένας ομιλητής, ο Παύλο Ρανζέλ. Και έχω μετά άλλους τέσσερις ομιλητές, αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, ας μου το πει τώρα γιατί πρέπει να ε, κανονίσουμε τον, ε, τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι εμένα δεν με ικανοποιεί τόσο πολύ όσο το συνάδελφο κ. Κόρμπετ η ιδέα ότι το Συμβούλιο τώρα θέλει να συμμετάσχει και να προσχωρήσει στην συμφωνία πλαίσιο. Ήμουν τελευταίο εισηγητή ε, αυτή τη συμφωνία πλαίσιο εδώ σε αυτή την επιτροπή. Και τότε επιμείναμε με πολύ έντονο τρόπο να υπάρχει συμμετοχή του Συμβουλίου στην, στην απόφαση, συμφωνία πλαίσιο συγγνώμη, και το Συμβούλιο αρνήθηκε. Μάλιστα, απείλησε και τα δύο θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο και Επιτροπή, με δικαστικές διαδικασίες, γιατί η απόφαση πλαίσιο υποτίθεται ότι ήταν παράνομη. Τούτου λεχθέντος πρέπει και εμείς να είμαστε ανοιχτή, να υπάρχει και παρουσία του Συμβουλίου, αλλά για τα ζητήματα που αφορούν μόνο τις ε, σχέσεις μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά λοιπόν, σε αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Γιατί μετά από αυτή την εξαιρετικά έντονη εμπειρία με τις ε, σχέσεις μας με το Συμβούλιο, γιατί τα γνώριζε όλα αυτό το Συμβούλιο, η πείρα μου λοιπόν μου δείχνει ότι ε, το Συμβούλιο τώρα θέλει να συμμετάσχει γιατί όταν, εφόσον δεν μπορεί να κερδίσει, θέλει να συμμετάσχει. Για να αλλάξει σημαντικά επιτεύγματα που έχουμε για την εισαγωγή και της διάστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Θετικέ λοιπόν οι εξελίξει, αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Γιατί εξαρτάται από το σχεδιασμό, το στόχο του Συμβουλίου. Τι θέλει το Συμβούλιο, καλύτερες διοργανικές ε, σχέσεις, τότε με τα χαράς. Αν θέλει όμως να προσπαθήσει να μειώσει την επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι θετικό. Επίσης, δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση του κυρίου Κόρμπετ για τη διαδικασία κίτρινης και πορτοκαλί κάρτας. Τώρα θα πρέπει να υπερασπιστώ την άλλη πλευρά από τη δική μου πείρα και εγώ συμμετείχα ενεργά και δραστήρια με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία πέντε χρόνια και βλέπω ότι αυτοί οι δύο μηχανισμοί δεν είναι αρκετά ευέλικτοι. Οι κυβερνήσεις έχουν λόγο να έχουν ένα τέτοιο αποδοτικό μηχανισμό κίτρινης και πορτοκαλί κάρτας και εγώ θα καταβάλω προσπάθειες να έχουμε καλή και εύρυθμη λειτουργία αυτών των δύο μηχανισμών πριν περάσουμε στην κόκκινη κάρτα. Οι κανόνες μας δεν είναι αρκετοί ευέλικτοι για να πάρει ικανοποιητικές διαστάσεις αυτός ο μηχανισμός. Και όταν δεν έχουμε πορτοκαλί και μόνο κίτρινες κάρτες, έχουμε δει μέχρι τώρα, σε 4-8 εβδομάδες είναι πολύ δύσκολο να βρούμε, να έρθουμε σε επαφή με όλα τα κοινοβούλια. Πρέπει λοιπόν να ε, δουλέψουμε με αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι καλά, και να τα κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά. Τέλος. πριν προσπαθήσουμε να παρέμβουμε στην απόφαση, στη συμφωνία πλαίσιο ε, μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, πρώτα θα πρέπει να περάσουμε στην ε, διοργανική ε, συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Είναι κάτι το οποίο αφορά και τα τρία θεσμικά όργανα και όπου μπορούμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Φυσικό και επόμενο είναι ότι κάποιες διατάξεις της ε, υφιστάμενης συμφωνίας πλαίσιο θα πρέπει ε, να μεταφερθούν στην συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Μάλλον. Αλλά αυτή την προσέγγιση θα προτιμούσα ως ε, μέλος του Κοινοβουλίου που επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση ε, του Κοινοβουλίου και των Ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Αυτές τις παρατηρήσεις έχω. Παρεπιπτόντως, νομίζω ότι δεν είναι πολύ καλό να έχουμε τους επιτρόπους στα Εθνικά Κοινοβούλια. Η Επιτροπή θα πρέπει να λογοδοτεί ενώ, ενώπιον ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικές κυβερνήσεις ενώπιον των Εθνικών Κοινοβουλίων. Στο, στα ομοσπονδιακά συστήματα δεν έχουμε τέτοια εμπειρία παρουσίας των μελών των εθνικών κυβερνήσεων στα κρατικά κοινοβούλια των επομένων των μελών. Δεν είναι αυτό συνήθι πρακτική. Και θεωρώ και λάθος να γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί τότε ε, να μειώνεται ο ρόλος και η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τον Υπουργό, απλώς για να ξεκινήσει μια συζήτηση με τους συναδέλφους. Ε, thank ε, you. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα έξι αγορητέ. Ε, παρακαλώ πολύ λοιπόν να μην ξεπεράσετε τα τρία λεπτά ο καθένας, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα μετά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως ε, με τα όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και όχι ιδεαλιστές. Δεν συμφωνώ με την άποψη η οποία λέει ε, ότι ε, οι αρχές της στήριξης και της βοήθειας εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο. Πιστεύω ότι μπορούμε ε, καλύτερα να ε, βοηθήσουμε την υλοποίηση από τεχνικά Κοινοβούλια. Η υπερβολική ε, νομοθέτηση νομίζω ότι δεν βοηθάει κανέναν. Ε, υπάρχει μία υπερπαραγωγή δικαίου, υπάρχει ε, ένας πληθωρισμός ε, νομοθετημάτων που δεν ικανοποιεί κανέναν. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να σταματήσει η υπερβολική νομοθέτηση. Τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η υπερβολικά ε, κεντρική ας πούμε διακυβέρνηση και πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, να τα δούμε αυτά με καθαρό βλέμμα. Εσείς ε, μιλάτε από την πλευρά του Συμβουλίου. Ε, θα πρέπει να δούμε με ποιο ορθολογικό τρόπο, με ποια πρακτικά μέτρα μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την υπερπαραγωγή νομοθεσίας. Ο κίνδυνος στο παρόν σύστημα είναι να βρούμε λύσεις ε, οι οποίες στην ουσία ε, οδηγούν στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ε, και βεβαίως εγώ ξέρω, ίσως δεν ξέρω τα πάντα όσον αφορά τις, τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ξέρω ποια είναι η συνταγή για μια καλή ευρωπαϊκή διαδικασία και ε, τα εθνικά κοινοβούλια ε, παραπονιούνται πολλές φορές ε, γιατί η αρχή της αλληλεγγύης δεν εφαρμόζεται με το σωστό τρόπο και άρα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τον μπούσουλα κατά κάποιο τρόπο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αποσύρει ορισμένα μέτρα όσον αφορά την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών που έδειξε ο κύριος Σέφλινγκ αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να εφαρμοστεί με καλύτερο τρόπο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι στην πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απορρίπτει και πρωτοβουλίες ε, οι οποίες ε, έχουν υπογραφεί από εκατομμύρια πολίτες. Εάν αυτές οι πρωτοβουλίες λοιπόν δεν ληφθούν υπόψη, αυτό θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο τους πολίτες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν με καλή πίστη ε, το δίκαιο και την νομοθεσία, τα θεσμικά όργανα. Εάν δεν έχουμε, αν δεν αποκτήσουμε μία ε, θετική ε, κουλτούρα, ας πούμε, θετική νοοτροπία, τότε πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα σταματήσουν να έχουν εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα επικεντρωθούν μονάχα στα εθνικά τους κοινοβούλια και δεν θα τους ενδιαφέρει πλέον τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είμαστε ευρωρεαλιστές. Κύριε Υπουργέ, α, κατά τη δική σας άποψη, ποιος θα ήταν ο μηχανισμός αυτός ο οποίος θα έδινε την δυνατότητα να σταματήσει αυτή, αυτός ο αυξανόμενος κεντρισμός. Thank you, Chair. Mr. Minister, you made... Ευχαριστώ κύριε κυρία Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στις κοινωνικές ρήτρες και αυτό με ικανοποιεί. Κατά την άποψή μου, περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη κοινωνική Ευρώπη, γιατί εάν ε, δυναμητήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό ε, μοντέλο, τότε δεν ε, θα υπάρξει καμία δυνατότητα να προσεγγίσουμε αυτό το μοντέλο το ευρωπαϊκό. Ε, η οικονομική διακυβέρνηση, πώς τη βλέπετε, κυρίως όσο και, τα μέτρα τα οποία αφορούν ε, την ε, διακυβέρνηση και την εφαρμογή της, πώς τα βλέπετε. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη, υπάρχει μεγάλη ανισότητα στις κοινωνίες μας και επίσης τα προγράμματα λιτότητας. Ποια άποψη έχετε για αυτά. Ξέρετε ότι προκαλούν ακραία κοινωνική μιζέρια, κυρίως στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την ε, συντομία σας, η Mercedes Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον ε, ε, Υπουργό Γκότσι ο οποίος ε, μας είπε ότι το θέμα των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν είναι ταμπού ε, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ίσως δεν ισχύει για όλες τις πρωτεύουσες, αλλά πάντως είναι ένα καλό νέο. Βεβαίως θα ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς εννοείται λέγοντας θεσμικά όργανα. Ενδεχομένως είναι και κάποια νέα συνθήκη όσον αφορά καλά στοχευμένα μέτρα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν από κοινού ας πούμε τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων, αυτή η αρχή της επικουρικότητας. Εγώ πιστεύω ότι μία από τις προτάσεις που κάνατε κι εσείς ο ίδιος και που ε, τελικά φάνηκε και στις παρεμβάσεις μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι δηλαδή ε, το να ζητήσετε, όχι να επιβάλλετε, να ζητήσετε από τους ε, υπουργούς ή από τους υφυπουργού, όσους τέλος πάντων είναι υπεύθυνοι για το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, να πληροφορούν εκ των προτέρων τα Εθνικά Κοινοβούλια για τα κεντρικά νομοθετικά θέματα, κυρίως όσον αφορά ας πούμε την, ε, τον νομοθετικό προγραμματισμό. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορούν να υπάρξουν ε, συναντήσεις ε, με τις νομοθετικές επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων όπου θα μπορούν να συζητιούνται από κοινού τα ζητήματα του νομοθετικού προγραμματισμού και επομένως να υπάρξει εκ των προτέρων διαβούλευση για όλα τα υποσυζήτηση ζητήματα. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο γιατί ε, και... Νομίζω ότι αυτή η δυνατότητα παρακολούθησης ε, της ε, συζήτησης και μια διαδικασία early warning ε, έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης, όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών, ξέρετε ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της ε, ε, Λισαβόνας μπορεί να προσφύγει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπώντας το υποπεριφερειακό επίπεδο. Αλλά ξέρω από την εμπειρία μου ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί στην πραγματικότητα είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα πλήρης ε, των κρατών ή πλήρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις αυτές. Στις, στις περισσότερες ε, φορές υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας. Επομένως, ο καθένας ε, υλοποιεί ένα κομμάτι της νομοθεσίας ενώ στο επίπεδο της δικιάς του αρμοδιότητας. Και αυτό ισχύει και για την διακυβέρνηση και σε πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης κτλ. Επομένως, τις περισσότερες φορές ε, δεν παραβιάζεται η επικουρικότητα αλλά η αναλογικότητα και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουλέψουμε. Είναι σπάνια η περίπτωση που κάτι μπορεί να κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μόνο η Κεντρική Κυβέρνηση ή μόνο η Περιφερειακή κυβέρνηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε ε, πολλές ε, περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, μπαίνει λίγο στα χωράφια, περισσότερο από όσο θα έπρεπε, στα χωράφια είτε της κεντρικής αλλά περισσότερο της περιφερειακής διακυβέρνησης και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε η αρχή της αναλογικότητας εγγενώς να περιλαμβάνεται στην αρχή της επικουρικότητας γιατί διαφορετικά ε, σας λέω δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσφύγει κανείς εναντίον της επικουρικότητας γιατί στην ουσία πρόκειται πάντα για αναλογικότητα. Επομένως αυτό που παραβιάζεται συνήθως είναι η αρχή τη αναλογικότητα και ουχή αυτή της επικουρικότητας. Και αυτό σα το λέω ε, γιατί τα έχω δει από την Επιτροπή των Περιφερειών πάρα πολύ συχνά τα έχω δει από μέσα. Και πολύ συχνά έχουμε ζημία ε, στο, των εθνικών, συγγνώμη, των, υπο, το, νομικών συστημάτων σε υποεθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και εκεί υπάρχει παραβίαση όχι της επικουρικότητας αλλά της αναλογικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ <clears throat> κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση του. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο θέμα του ελέγχου της επικουρικότητας και της λεγόμενης κίτρινης κάρτας. Με εκπλήσει λιγάκι το ότι είπατε ότι <clears throat> πάρα πολλοί θεωρούν ότι λειτουργεί καλά αυτός ο έλεγχος επικουρικότητας γιατί χρησιμοποιήθηκε μόνο δύο φορές τα τελευταία πέντε χρόνια για να, να επιτευχθεί ο αριθμός των κοινοβουλίων που ξεκινάει τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό γίνεται... γιατί η Κομισιό δεν κάνει ποτέ σφάλματα ή αλλιώς μπορεί κανείς να θέσει το ερώτημα μήπως γίνεται αυτό επειδή τα εθνικά κοινοβούλια έχουν διαφορετικούς βαθμούς φιλοδοξίας. Πόση ενέργεια, πόση δουλειά θέλουν να επενδύσουν σε αυτή την υπόθεση του ελέγχου της ε, επικουρικότητας. Αυτό είναι κάτι που ποικίλει πολύ από χώρα σε χώρα. Όταν δούμε τις στατιστικές σε σχέση με αυτές τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία της κίτρινης κάρτας, βλέπουμε ότι είναι πολύ μορφή η κατάσταση, πολύ διαφορετική από κράτος μέρος σε άλλο. Για να λειτουργήσει λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα, Θα πρέπει η διαδικασία της κίτρινης κάρτας να είναι απλούστερη. Και αναρωτιέμαι αν πρέπει να έχουμε πράγματι 8 εβδομάδες περιθώριο και το 1 τρίτο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μπορούμε με καλύτερο συντονισμό να βελτιώσουμε αυτή τη διαδικασία. Προς το παρόν, εγώ δεν βρίσκω ικανοποιητική αυτή τη διαδικασία. Thank you. Ε. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Υπουργό για την παρουσίαση. Δύο σύντομες ερωτήσεις, ε, γιατί ε, άλλες έχουν ήδη υποβληθεί. Η πρώτη αφορά τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήθελα να ρωτήσω μήπως σκόπιμο θα ήταν να περάσουμε από έναν ρόλο ουσιαστικά αρνητικό, δηλαδή την δυνατότητα άσκησης βέτο, ε, ε, να φτάσουμε ε, σε δύο θέματα όσον αφορά δηλαδή το θέμα της, ε, των οικονομικών προοπτικών και όσον αφορά το θέμα της ε, συνταγματικής αναθεώρησης σε μια θετική διαδικασία. Ε, σας το λέω γιατί εσείς γνωρίζετε το θέμα ε, των κοινοβουλευτικών διασκέψεων, των ΑΣΥΖ για για το μέλλον της Ευρώπης. Έχετε λοιπόν κάτι να πείτε σε σχέση με αυτό. Δεύτερον, πολύ σύντομη ερώτηση γιατί έχει ήδη υποβληθεί. Λέτε κύριε Υπουργέ ότι για το μέλλον ε, των, ε, για το μέλλον των θεσμικών οργάνων βρήκατε ευνοϊκότερο κλίμα ε, σε εθνικό επίπεδο ευνοϊκότερο κλίμα λοιπόν στις πρωτεύουσες από ό,τι στις Βρυξέλλες. Τι εννοείται ευνοϊκότερο κλίμα? Ευχαριστώ. Ο κύριος Πλάκοβιτς, τελευταίος ομιλητής. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Χούμπνερ. Καλημέρα Σάντρο. Όπως και πολλοί συνάδελφοι ε, ανέφεραν πολλά σημαντικά θέματα, θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα βεβαίως να σε ευχαριστήσω για το briefing ε, το οποίο μας έκανε όσον αφορά και την άτυπη ε, διάσκεψη του Μιλάνου. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω, που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον δηλαδή να μάθω, τώρα που ε, θα έχουμε τον κύριο Τίμερμανς υπεύθυνο για τις διοργανικές σχέσεις. Είδαμε στην περίπτωση της Κόζακ όπου οι Ολλανδοί συνάδελφοι πάντα προωθούν το επιχείρημα, προτάσουν το επιχείρημα ότι η Ευρώπη πρέπει να υπάρχει εκεί που είναι απαραίτητη. Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως ε, ο αντίκτυπος ε, του δημοψηφίσματος του 2005 και το διαπιστώνουμε αυτό όταν μιλούν οι Ολλανδοί συνάδελφοι. Εσείς σαν υπουργό είπατε ότι δεν θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις σε σχέση με τη Λισαβόνα. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το μήνυμα στα πλαίσια μιας ευρύτερη συζήτησης για την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ε, αυτή τη έννοια τη αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω και στον Ρίτσορτ Κόρμπετ, έστω και αν ε, δεν είναι ε, εδώ. Συνήθω δεν απαντώ σε αυτού που κάνουν μια ερώτηση και φεύγουν, αλλά επειδή τα εξήγησε πολύ καλά θα ήθελα να το απαντήσω. Έλεγε λοιπόν ο κύριο Κόρμπετ ότι πρώτα απ' όλα το θέμα του κατά πόσον ε, ε, ε, πρέπει ή θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να ακούω τις απόψεις, μας γι αυτό, απόψεις σας, μα γι' αυτό είμαι εδώ, για να τις ακούσω και θα προσπαθήσω να τις αποθυσαυρίσω και να τις χρησιμοποιήσω όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό επιδιδόμαστε αυτή την άσκηση. Όσον αφορά τη συμφωνία πλαίσιο, την οποία ανέθιξε ο συνάδελφος Κόρμπετ, αλλά και ε, και ο, ο κύριος Ράντζελ είπα είπα στην αρχική μου τοποθέτηση ότι ως ε, ε, Προεδρία θεωρούμε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει με προσοχή το ενδεχόμενο να υποβάλει στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο το θέμα της συμφωνίας αυτής είναι γεγονός ε, και το είπα και αυτό ότι μια και μπαίνουμε σε μια νέα φάση θα πρέπει να συζητηθούν και κάποιες άλλες απόψεις ενδεχομένως ε, να ενδυναμώσουμε όπως έλεγε άλλωστε και ο Σανφο Ρανζέλ ορισμένα πράγματα και ενώ μεταξύ αξιολογούμε εάν όλες ε, οι αντιπροσωπείες θα συμφωνήσουν με την, με την άποψη που εκφράζει η Προεδρία. Οι Άγγλοι λένε η take two του τάγκο αλλά εδώ ακόμα και για αυτό το περίφημο ταγκό τρεις χρειάζονται. Επομένως θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να χορέψουμε στο τέλος κατά τη δικιά μου άποψη καλύτερα θα ήταν να επιστρέψουμε στην ιδέα της καλής συνεργασίας μεταξύ των τριών και όχι ε, να κάνουμε ειδικέ σχέσεις ανά δύο. Μία ιδιαίτερη σχέση Κομισιόν-Κοινοβούλιο, μία άλλη ειδική σχέση ε, Συμβούλιο-Κομισιόν. Ε, κατά τη δική μου άποψη χρησιμότερο θα ήταν να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε και οι τρεις άλλωστε. Τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των ε, ε, πολιτών. Είναι τρία τα θεσμικά όργανα τα οποία θα πρέπει ε, να συνεργάζονται έτσι ώστε να φτάνουμε σε πολιτικά συμπεράσματα και σε πολιτικές πράξεις. Δεν είναι δύο ξεχωριστά και γι' αυτό λοιπόν θέσαμε πρώτο το ζήτημα αυτό γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων να εξυπηρετεί τους σκοπούς και στόχους που θα έχουν ταυτοποιήσει ως στρατηγικούς στόχους, ως επιχειρησιακούς στόχους το Συμβούλιο, ε, η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να δούμε ε, επομένως και δεν θέλω να μπω εδώ στις πολιτικές δυναμικές εγώ δεν θέλω να παρέμβω στις, στους, στις συμφωνίες ή τις ισορροπίες μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών απλώς εμείς θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος, ας πούμε, ε, κύριος Γιούγκερ ε, προετοίμασε τα διάφορα χαρτοφυλάκια και τις, ε, τη, τη, τη, λειτουργία της Κομισιόν, θεωρούμε ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί πραγματικά έχει λάβει υπόψη τους στρατηγικούς στόχους. Είναι μια προσέγγιση που κατά την άποψή μας θα πρέπει γενικώ να ακολουθούμε. Επίσης και ο κύριος Κόρμπετ και άλλοι αναφέρθηκαν και η κυρία Μπρέσο και ο κύριος Κόρμπετ και ο κύριος Άντερσον αναφέρθηκαν στο θέμα της επικουρικότητας και στο θέμα της ε, λειτουργίας της. Έχω να πω αρκετά πάνω σε αυτό. Δεν είπα, ε, συνάδελφε Άντερσον, ότι όλα λειτουργούν σωστά ε, στον τρόπο με τον οποίο ε, υλοποιούνται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Είπα ότι υπό το φως των εργασιών που έχουν ξεκινήσει το Συμβούλιο, οι αντιπροσωπείες και τα κράτη-μέλη φρονούν ότι δεν είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε να βελτιωθεί η υλοποίηση αυτών των δύο αρχών. Είναι διαφορετικό λοιπόν. Ε, όμως συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε και αυτά που είπε και η κυρία Μπρέσο όταν στην ουσία ε, είπατε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα εθνικά κοινοβούλια ε, και οι ε, τοπικές αυτοδιοίκησεις χρησιμοποιούν ή αντιμετωπίζονται σε σχέση με τις δύο αυτές αρχές και επομένως ε, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που είπε η συνάδελφος Μπρέσο όταν ε, είπε ότι έννοια έχει όλη αυτή η διαδικασία εάν δούμε ακριβώς πώς ε, υλοποιούνται και η αναλογικότητα και η επικουρικότητα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι στο δικό μου Εθνικό Κοινοβούλιο ήρθα σε αντίθεση με πολλούς γιατί το Κοινοβούλιο μου έλεγε ότι όχι, όχι, θα μιλήσουμε μόνο για επικουρικότητα και όχι για αναλογικότητα. Και ε, ε, εγώ είπα ότι ε, θα πρέπει να δούμε καλύτερα. Δεν μπορεί μονάχα να ελέγχει το Εθνικό Κοινοβούλιο την ακριβή υλοποίηση της επικουρικότητας, γιατί όπως είπε και η Στράνθος Μπρέσο, πολλά προβλήματα σχετίζονται με την αναλογικότητα και όχι με την επικουρικότητα και ε, επομένως, ε, ωστόσο πρέπει να πω ότι ότι περισσότερο εξαρτάται αυτό από το πώς ερμηνεύουν τις αρχές αυτές τα εθνικά κοινοβούλια και πόσο ε, θέλουν, σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Εξαρτάται περισσότερο από αυτούς παρά από την άλλη πλευρά. Παρόλα αυτά, οπωσδήποτε πολλά μπορούν να βελτιωθούν στις σχέσεις μεταξύ Κομισιών και Εθνικών Κοινοβουλίων και οπωσδήποτε χρήσιμο είναι ε, να χρησιμοποιηθεί η ΚΟΖΑΚ ακριβώς, η οποία είναι αρμόδια επί της ε, ουσίας για να συζητηθούν τα θέματα αυτό και ε, χρήσιμο θα ήταν να συζητάτε τα θέματα αυτά στην ΚΟΖΑΚ με τους συναδέλφους σας των άλλων εθνικών κοινοβουλίων. Μερικοί μεταξύ ημών είπατε και επιστρέφω ξανά και σε ερώτηση που υπέβαλε ο κύριος Κόρμπετ, ότι εξαρτάται πολύ από τις σχέσεις ανάμεσα στην ε, Εθνική Κυβέρνηση και το Εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι μια συζήτηση την οποία έχουμε ξανακάνει στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε, είπαμε ότι η κάθε κυβέρνηση, το κάθε εθνικό κοινοβούλιο οργανώνεται όπως θέλει. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Ε, ε, εμείς στην Ιταλία εγκρίναμε ε, το 2012 μια, ένα νόμο ο οποίος πολύ βελτιώνει τις σχέσεις ανάμεσα ε, στο κοινοβούλιο και την ε, κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως κάποια κοινοβούλια που δεν θέλουν. Ε, επίσης πρέπει να σας πω ότι η Προεδρία δεν έχει κανένα πρόβλημα με την φράση «ever closer union» Ε, απλώς εμείς λέμε ότι δεν θα υποβάλουμε το ζήτημα αυτό ε, σε συζήτηση. Εμείς δεν θέλουμε όμως να διαγραφεί αυτή η φράση Ever Closer Union. Ε, Σάλφο Σέφλινγκ αναφέρθηκε ο συνάδελφος στην πρωτοβουλία ή μάλλον όχι. Να σας πω ότι ήδη απάντησα σε ορισμένα από τα σχόλιά σας, αλλά αναφερθήκατε στην ε, ανάγκη αναθεώρησης της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν λειτουργήσε πάρα πολύ καλά αυτή η πρωτοβουλία. Θα πρέπει από κοινού να εργαστούμε έτσι ώστε να δούμε πόσο από την, πόσο κομμάτι από αυτή την κακή λειτουργία αφορά την Κομισιόν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το, την πρωτοβουλία των πολιτών ε, το Ευρω... διορθώνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, πόσο είναι πρόβλημα εγγενές της ίδιας της μορφής της πρωτοβουλίας ή αν είναι πρόβλημα κρατών μελών. Πόσο υλοποίησαν ας πούμε και η ε, πρωτοβου... πόσο υλοποιήθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Ο τρόπος π.χ. συλλογή των ε, υπογραφών με ηλεκτρονικό τρόπο, με μη ηλεκτρονικό τρόπο κτλ. Υπάρχουν μία σειρά πράγματα τα οποία θα πρέπει να ε, τα ξαναδούμε. Και αυτή είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση πρωτοβουλία η οποία έχει τεράστιο δυναμικό, το οποίο ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί και οπωσδήποτε αυτό το σημείο θα συζητηθεί ξανά στα πλαίσια των εργασιών μα και οπωσδήποτε στην τελική μα έκθεση θα το αναφέρουμε. Στον συνάδελφο Ζολάινεν μπορώ να πω το εξή. συνεργαζόμαστε όχι μονάχα στα πλαίσια της Προεδρίας αλλά και ο Πρωθυπουργό Ρέντσι το είπε όταν μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη more or less Europe το θέμα είναι να έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη better Europe σας το είπε και το πιστεύουμε αυτό. Πρέπει να ε, βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή δράση απλουστεύοντας την πρώτα απ' όλα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί ε, και οπωσδήποτε θα πρέπει να ξαναδούμε το νέο τρόπο υλοποίησης, εφαρμογής των παλαιών αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο γίνεται, υλοποιείται η Ευρώπη. Ε, γιατί μερικές φορές είναι πολύ ε, ε, περιγραφική, μερικές φορές μπαίνει σε υπερβολικές λεπτομέρειες, άλλες φορές δεν μπαίνει σε αρκετές λεπτομέρειες και δεν δίνει αρκετές ενδείξεις. Θα πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Τώρα, το θέμα των αποφάσεων, αν θα πρέπει να παίρνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία κτλ. είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στην άτυπη διυπουργική του Μιλάνου. Ε, εφήγει και οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει, όπως θα μας απασχολήσει άλλωστε και ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα ε, έχει χρησιμοποιηθεί η ενισχυμένη εργασία. Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι και οι Πασερέλ και οι ενισχυμένες συνεργασίες είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και ε, ε, πρέπει να πω ότι εξαρτόμαστε και από τον τρόπο υλοποίησης αυτών των μέτρων αλλά κυρίως εξαρτόμαστε από την πολιτική βούληση να τα ε, υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά ήδη στον συνάδελφο Ραντζέλ όσον αφορά την, ε, ε, καλύτερη, το καλύτερα νομοθετήν. Ναι, συμφωνούμε κύριε Ραντζέλ και είμαστε πολύ ανοιχτοί ε, και νομίζω απλώς ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πεποίθηση, μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, μεγαλύτερη πίστη στα αυτά που λέμε, να δούμε ενδεχομένως και να ξαναδούμε κάποια, σημεία τη συμφωνίας πλαίσιο Κοινοβουλίου Κομισιόν Στον κύριο Ζοντόφσκι να πω, να τον, ε, διασφα... Ε, να, να τον ε, του πω ότι δεν μίλησα νομίζω με έτσι, πνεύμα ιδεαλιστικό. Ιδεο... Νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ πραγματιστής και φυσικά συμφωνώ ότι θα πρέπει η προσέγγιση να είναι απτή, πραγματιστική, ορθολογική, συγκεκριμένη και με αυτόν τον τρόπο νομίζω προσεγγίσαμε τα πράγματα γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε καλύτερα να υπηρετήσουμε και τους στόχους μας αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Κύριε Κατρούγαλε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ε, την παρέμβασή σας για τα άρθρα 8 και 9 και χαίρομαι ε, που σήμερα ε, αξιολογείται θετικά το ότι το ζήτημα έχει αρχίσει και συζητιέται, έχει μπει στο τραπέζι. Βρίσκεται στο τραπέζι λοιπόν το θέμα ε, και της, ε, ε, και της ανεργίας και της απασχόλησης και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και για μας. Πρόκειται για μια εργασία πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι αντιστάσεις είναι πάρα πολλές. Αντιστάσεις στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων για να αντιμετωπιστεί ακόμα ευρύτερα το ζήτημα, δηλαδή το πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτή η στόχοι που βρίσκονται πλέον στο ε, τραπέζι και που τα συζητάει η ομάδα ε, των φίλων της Προεδρίας, αλλά εσείς πήγατε και πιο μακριά και συμφωνώ μαζί σας. Λέτε, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, εξελίξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ γρήγορες στα πλαίσια της οικονομικής governance, της οικονομικής διακυβέρνησης, δεν θα πρέπει να δούμε κατά πόσον σωστά ή λάθος έχουν προσαρμοστεί οι πολιτικές ε, οι πολιτικές σε αυτές τις νέες συνθήκες. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και το συμμερίζομαι απολύτως, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αντιστάσεις και δεν εγώ πιστεύω, πιστεύω πάρα πολύ στα θέματα αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί ε, και σε πολιτικό επίπεδο συμφωνία. Γι' αυτό θα το επανυποβάλλω. Ε, κάτι άλλο το οποίο με ρωτήσατε ε, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τον ε, στόχο της συνάντησής μας. Αλλά δράτω με τις ευκαιρίες για να σας πω ότι η, διαδρομή μας είναι αρκετά σαφής. Τον Ιούνιο οι, αρχικές, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αυτή στην ατζέντα Βαν Ρομπόη και συζητώντας την ε, είπαν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο η ευελιξία η οποία υπάρχει στις ε, συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει σταθερότητα στην ανάπτυξη. Ε, ε, εκεί υπόθηκε λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί όθηση στην πολιτική των επενδύσεων και στην ανάπτυξη. Εμείς σαν ε, Ιταλία, σαν Προεδρεύουσα, κάναμε κάποιες κινήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι η ατζέντα του Προέδρου Γιούγκερ είναι μια χρήσιμη ατζέντα και περιμένουμε πλέον η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκμεταλλευτεί την στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ευελιξία την οποία παρέχουν ε, οι συνθήκες. Ήταν σαφής ο τρόπος με τον οποίο και βάσει ποιου σκεπτικού οι 28 ε, ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επέλεξαν τον ε, πρόεδρο Γιούγκερ. Ήταν σαφές ότι θα γίνει μια προσπάθεια εξέβρεσης και επιπλέον πόρων. Αυτό ήταν σαφές από την αρχή και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε και κάποιες πιο θετικές συγκεκριμένες απτές ενδείξεις στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για να δούμε ποιο δρόμο ε, ε, ε, ακολουθεί τελικά η Επιτροπή. Στην συνάδελφο Σπινέλη εγώ στην τελευταία συνεδρίαση ε, είχα επιβεβαιώσει τον φεντεραλισμό μου όχι σαν εκπρόσωπος της προεδρεύουσας χώρας αλλά ε, σαν Ευρωπαίος πολίτης. Το επαναλαμβάνω και το επιβεβαιώνω και θεωρώ ότι το θέμα των ασίζ, των κοινοβουλευτικών ασίζ, το θέμα ε, της όθησης που θα πρέπει να έρθει από τα εθνικά κοινοβούλια είναι μια πολύ καλή ιδέα. Είναι μια ιδέα βάσει της οποίας τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συνεχίσουν τις σκέψεις, ε, τις σκέψεις τους. Και εσείς, όπως και η συνάδελφος Μπρέσο, ε, έθιξαν λίγο το ζήτημα αυτό των ε, πρωτευουσών και της αντιμετώπισης που την χάνει το θέμα της αναθεώρησης των συνθήκων στις ε, πρωτεύουσες. Ε, κοιτάξτε, υπάρχει μία πρώτη συμφωνία έτσι ώστε να ξεκινήσει, όπως και ξεκίνησε, η ε, δουλειά όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για να δούμε στο εσωτερικό της συνθήκης της Λισαβόνας τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα, εγώ δεν μπορώ να εκφράσω εδώ τη θέση της Προεδρίας, την προσωπική μου θέση μπορώ να σας πω, ότι εάν η νέα Εάν, στην νέα ε, κοινοβουλευτική ε, εντολή καλό θα ήταν ε, να δούμε ενδεχομένως και το θέμα της αναθεώρησης των συνθήκων όπως με ρώτησε η κυρία Μπρέσο, εγώ είμαι θετικά διακείμενος αλλά είναι η προσωπική μου άποψη, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου, είναι η δικιά μου άποψη σαν εκπροσώπου, σαν μέλους της Ιταλικής κυβερνήσεως. Τώρα, κατά πόσο είναι ταμπού το ζήτημα αυτό, τι να σας πω. Είπα και προηγουμένως και το ξαναλέω, ότι κοπιάσαμε περισσότερο να πείσουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την καλή πίστη της προσπάθειάς μας παρότι δουλεύουμε βάσει συγκεκριμένων νομοθετικών ε, ε, κειμένων, τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι, περισσότερο στις Βρυξέλλες και λιγότερο στις πρωτεύουσες, υπάρχουν πολλοί λοιπόν που θεωρούν ότι... Ε, το να συζητάμε για τα, για θεσμικά όργανα τη στιγμή που έχουμε τόσα σημαντικά πράγματα να πούμε γίνεται λίγο δευτερεύον για την ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Ε, η δικιά μου προσωπική θέση ε, δεν είναι καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Αγαπητές, Γένκοβιτς, σας ξέρω από την ε, υπερπεριφέρεια Ιωνίου Αδριατικής ε, και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Ε, πρέπει να σας πω ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ήταν πολύ ανοιχτό, πολύ δεσμευμένο ε, δεν ακούσαμε από τον Φρανς Τίμερμανς σαν εκπρόσωπο της Ολλανδικής κυβέρνησης ε, να έχει διάθεση συγκράτησης της διαδικασίας ή παρεμπόδισης. Κοιτάξτε, εγώ, εγώ ε, είδα τον Φραντ Τίμερμανς να έχει ε, έτσι πολύ, να είναι πολύ πεπισμένο σαν μέλο τη ε, Ολλανδικής Αντιπροσωπείας ε, και το θέμα της θεσμικής μεταρρύθμιση είναι ένα θέμα τον οποίο τον απασχολεί πάρα πολύ μαζί με την ασφάλεια, μαζί με τη διακυβέρνηση, μαζί με την συνταγματική και νομοθετική σταθερότητα και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι και η Vivian Redding έκανε πάρα πολύ θετικά πράγματα και η γενική μας αξιολόγηση είναι θετική όσον αφορά την ε, διαθεσμική συνεργασία. Και, και ο κύριος Τίντερμανς ε, κατέδειξε την σημασία που θα πρέπει τα θέματα αυτά να έχουν στη νέα ε, κοινοβουλευτική θητεία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό εξ ονόματός σας και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία γιατί νομίζω ότι τα συμπεράσματα των εργασιών αυτής της ομάδας, των φίλων της Προεδρίας και του Συμβουλίου μπορούν να είναι σημαντικά στοιχεία για το δικό μας πρόγραμμα επίσης ως Συνταγματικής Επιτροπής. Και τώρα Περνάμε στο επόμενο σημείο της μέσης της διάταξης που είναι η, συζητή, η συζήτηση με εμπειρογνώμονες για τις θεσμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε υπήρξαν συζητήσεις και μεταξύ των συντονιστών για να προετοιμάσουμε μια απόφαση για το πρόγραμμα εργασίας μας για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το θεσμικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες σήμερα ενώπιόν μας που τους ζητήσαμε να μας παρουσιάσουν την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από θεσμική έποψη. Να έχουμε λοιπόν και τη δική τους αρρωγή με διαφορετικές οπτικές γωνίες και να μας πούν τι θεωρούν αυτοί ότι είναι οι προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι προκλήσεις θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των τωρινών συνθηκών και επίσης ποιες προκλήσεις θα είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν με τροποποίηση των συνθεκών και εισαγωγή νέων στοιχείων. Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σε αυτόν τον προβληματισμό για το πώς να χρησιμοποιήσουμε το τωρινό πλαίσιο. Τρεις εμπειρογνώμονες έχουμε. Το Γιάννη Μανουηλίδη, πολιτικός αναλυτής, αλλά και επικεφαλής του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής της Βρυξέλλες, ο Γιέκτε Φαν, ο οποίος είναι καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Εράσμιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο της Χάγης και είναι και Γενικός Γραμματέας της Διευρωπαϊκής Ένωσης Μελετών και ο Πρεσβευτής Δεσκουτέτε, ο οποίος για όλους εσάς που είσαστε παλιοσυρές είναι ένα σύμβολο της ε, διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο δρόμο για το 2004, ο πρέσβης Φιλίπ Τεσκουτέτε θα έρθει στη συνεδρίασή μας λίγο αργότερα, γιατί προς το παρόν δεν μπορεί να είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρότεινα λοιπόν να ακούσουμε πρώτα τους δύο εμπειρογνώμονες που είναι μαζί μας και στη συνέχεια μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση και μετά θα έρθει ο πρέσβης Δεσκουτέτα και θα έχει την ευκαιρία να λάβει το λόγο. Δεν θέλω από τους δυο σας θεωρείτε ότι πρέπει να λάβει πρώτος το λόγο. Ο Γιάννης, εντάξει. Γιάννης Εμμανουηλίδης. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. μεγάλη χαρά και είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας για να εξετάσουμε τις ε, Μελλοντικέ προκλήσεις σε θεσμικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα επόμενα 15 λεπτά θα ασχοληθώ με τα δύο αυτά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση για τα θεσμικά ζητήματα στην Ένωση, πρέπει να εξετάσουμε τα περαιτέρω στοιχεία πέραν ε, της, πέρα της τελευταίας ήταν ενδιαφέροντα αυτά τα τελευταία χρόνια, πρέπει να έχουμε λοιπόν κατά νου τα όσα συνέβησαν στον ε, τελευταίο πολιτικό κύκλο και τώρα να περάσουμε μετά και στις μελλοντικέ προβλέψεις. Ποιε θα μπορούσαν λοιπόν να είναι οι μελλοντικέ εξελίξει στο θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, για την ε, τρέχουσα κατάσταση σήμερα στην Ένωση είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να κάνουμε και προβλέψει για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, πέρασε από μία ε, θεμελιώδη κρίση, αν και δεν ήταν η χειρότερη από τις κρίσεις που είδαμε την τελευταία δεκαετία. Ελπίζω τώρα να με ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, ήταν μία πολύ σοβαρή κρίση, λοιπόν. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση ε, με αυτή την μεγάλη κρίση της Ευρωζώνης, ευρύτερη όπως επιλέξετε να την αποκαλέσετε. Πλέον βλέπουμε ότι έχουμε καλύτερους συστημικούς όρους σε σχέση με το 2012. Και λέω συστημικούς γιατί αν πείτε σε κάποιον ε, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το 2012, θα μα πούνε «Ε, πλάκα μα κάνετε. Ε, η δική μα εντύπωση δεν είναι ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, όμω από συστημική πλευρά έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, γιατί αυτό ο κίνδυνο να ξεφύγουν από τον έλεγχό μα τα πράγματα και να καταρρεύσει το ευρώ με όλες τις πιθανές επιπτώσεις αυτού του γεγονότος. Τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε ξεπεράσει συνολικά την κρίση. Δεν έχει περάσει η κρίση ούτε για αστείο και γενικά η οικονομική και πολιτική κατάσταση παραμένει ε, ασταθής και ευμετάβλητη και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κλιμάκωση στο μέλλον. Δεν λέμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά και όμως και χωρίς πιθανή κλιμάκωση υπάρχουν και σημαντικές ε, επιπτώσεις της κρίσης, οικονομικές, κοινωνικές, φορολογικές. Και όλα αυτά θα μας επιβαρύνουν και για τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι οι δύο στρατηγικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε είναι η πρόκληση του κατακαιρματισμού και η πρόκληση της απώλειας εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι ένα εγχείρημα που ε, ε, ωφελεί όλους. Καταγραμματισμό. Καταγραμματισμό μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτών. Οι πολίτε έχουν γυρίσει την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και οικονομικό καταγραμματισμό μεταξύ κρατών μελών που αυξάνεται. Καταγραμματισμό μεταξύ ε, κρατών μελών και εθνικών κοινωνιών. Στερεότυπα, μυσαλλοδοξία, όλα αυτά μπορεί να έχουν κορυφωθεί τώρα, αλλά νομίζουμε ότι θα παραμείνουν όλα αυτά στη συλλογική μνήμη των πολιτών. Κοινωνικό και πολιτικό κατακαιρματισμό μεταξύ κρατών μελών, δεν χρειάζεται να επισέλθω σε λεπτομέρειε. Υπάρχει ε, αυξανόμενος διχασμός μεταξύ των ε, πλουσιότερων και φτωχότερων των συλλογικών κρατών κατακαιρματισμό σε πολλούς τομείς λοιπόν και υπάρχει και αυτή η έλλειψη του win-win της, ε, των ωφελιών για όλους, για, για τα κράτη-μέλη, για όλους τους πολίτες. Υπάρχει η αίσθηση ότι πλέον δεν είναι ένα εγχείρημα που επωφελεί όλους, ότι το κόστος και τα κέρδη δεν ε, κατανέμονται ισότιμα. Υπάρχει φόβος ε, διάσπασης μεταξύ του πυρήνα και της περιφέρειας. Αν εξετάσετε τον προηγούμενο ε, πολιτικό κύκλο, υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις που αποτέλεσαν αντικείμενο και αποτέλεσμα ε, κάποιων θεσμικών ε, εξελίξεων, αλλά και ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων. Και θέλω να επικεντρωθώ σε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί συνδέονται και με τις θεσμικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω δύο κύριε, τρεις κύριες εξελίξεις που ήταν τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως η θέση σε ισχύ της συνθήκης της θα δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Μετά, από το 2010 έως το 2013 είδαμε ότι ήταν εξαιρετικές συνθήκες, έκτακτες συνθήκες. Περάσαμε την κρίση και ξέρετε ότι στην κρίση αναλαμβάνει ηγητικό ρόλο το εκτελεστικό σκέλος. Αυτό συμβαίνει πάντα και συνέβη και αυτή τη φορά. Δεν ε, πρέπει να σας εκπλήσει λοιπόν ότι η αρχική κρατών και κυβερνήσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διαδραμάτισαν τόσο σημαντικό ρόλο ε, στο θεσμικό σκηνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είχαμε έκτακτες περιστάσεις. Είδαμε ακόμα και ε, διακυβερνητικές συμφωνίε και εκτό του πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και μπορεί κάποιος ε, να τονίσει ότι ε, πρόκειται για αντίθεση μεταξύ του ευρωπαϊκού οράματος και του διακυβερνητικού μοντέλου. Και δεν θα έσφαλε κανείς να κάνει αυτή τη διαπίστωση. Υπάρχουν τέτοιες πρακτικές κατά τη διάρκεια μιας κρίσης αλλά δεν χρειάζεται να γενικεύουμε και να υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα τόσο εύκολα, γιατί ε, ακόμα και ε, ε, υπήρξαν αυτές οι διακυβερνητικές συμφωνίες, αλλά συμμετείχε και η Επιτροπή, υπήρχε και το Κοινοβούλιο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν μόνο διακυβερνητικό ε, φορέα, αλλά προσπάθησε να μεσολαβήσει. Λειτουργήσε, έδρασε και υπερεθνικά, λοιπόν. Δεν χρειάζεται να υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα. Υπάρχει μια τρίτη εξέλιξη, ένα φαινόμενο που έχουμε εντοπίσει και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε εδώ, που επηρέασε και το θεσμικό σκηνικό, μια ανισορροπία ή μάλλον μια νέα ισορροπία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου με κάποιες χώρες, ιδιαίτερα η πατρίδα μου, ε, η Γερμανία, ε, δεμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο και βλέπουμε ότι καμία απόφαση δεν, δεν μπορούσε να ληφθεί χωρίς τη Γερμανία, τη σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας. Αυτό συνδέεται με την ισχύ της Γερμανίας αλλά και με την έλλειψη ισχύω άλλων χωρών, ιδίως τη Γαλλία. Αυτό είναι κάτι καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τη Γερμανία που δεν έχει συνηθίσει να βρίσκεται έτσι ε, επικεφαλής. Βλέπουμε λοιπόν τον ε, ισχυρό ρόλο των κυβερνήσεων, πολιτική επιρροή του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και ισχυρός ρόλος της Γερμανίας έδωσαν όλα αυτά στην εντύπωση ότι δεν υπάρχει εξισορρόπηση των εθνικών συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια γενική εντύπωση που έχει επηρεάσει τους πάντες ε, την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Ο τελευταίος κύκλος πολιτικής λοιπόν ήταν εξαιρετικός, έκτακτος μάλλον. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε προς το που θα κινηθούμε, αλλά θα περάσουμε σε ένα νέο πρότυπο θεωρούμε και πλέον είναι ένα εγχείρημα, μια προσπάθεια να μαντέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον, με μια κρυστάλλινη σφαίρα. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να δώσουμε προγνωστικά για το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Φανταστείτε αν ήταν κάποιο πριν από πέντε χρόνια εδώ, στον τον, στην αρχή τη νέα ε, περίοδου, ποιο θα μπορούσε να φανταστεί τα όσα θα συνέβαιναν ε, την επόμενη πενταετία. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να κάνουμε κάτι αντίστοιχο τώρα, αλλά μπορώ να μοιραστώ μαζί σε κάποιες σκέψεις. Δύο είναι οι ενδιαφέρουσες εξελίξεις που ε, λειτουργούν μάλιστα και αντίθετα. Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που βλέπουμε να επιδρούν ταυτόχρονα. Πρώτον έχουμε μια αυξανόμενη πολιτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δείτε τώρα την ε, συζήτηση για την νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τις ακροάσεις, βλέπουμε ότι γίνεται πιο πολιτική η διαδικασία. Αυτό οφείλεται βεβαίως ε, στην αύξηση της προσωποποίησης και έχουμε και τους Spitzenkandidaten, τους ε, επικεφαλείς, τους κύριους υποψηφίους, ότι ο κύριος Γιούνκερ έγινε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά δείχνουν ότι γίνεται πιο προσωποπαγής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Βάιλερ τις αρχές της χρονιάς έλεγε ότι αυτό το καινοτόμο στοιχείο των Spitzenkandidaten μπορεί να είναι η πιο σημαντική από τις ε, νέες εξελίξεις που βλέπουμε στο πολιτικό επίπεδο. Αυτά μου έλεγε το Μάρτιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά βλέπουμε ότι είναι σημαντικές εξελίξεις. Η διαδικασία του, των candidate ήταν ένα ε, πείραμα που έγινε λίγο τσαπατσούλικα εντό αγωγικών. Ναι, οδήγησε σε αυτή τη διαδικασία η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά δεν είχε προγραμματιστεί έτσι. Όμω, βέβαια, αυτό αποτελεί τμήμα μια δυναμική διαδικασία. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την πρώτη εμπειρία που είχαμε το 2014. Θα αλλάξουν τα πράγματα το 2019, το 2024. Πρέπει όλοι να μάθουμε λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, τα πολιτικά κόμματα, οι κυβερνήσει, αλλά και τα μέσα μαζική ενημέρωση που διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο κατά την μεταφορά ε, των μηνυμάτων των ε, υποψηφίων προς το ευρύ κοινό. Αλλά θεωρώ ότι θα παραμείνει το πείραμα αυτό, αυτή η διαδικασία και δεν θα επανέλθουμε σε μυστικές διαπραγματεύσεις ε, πίσω από κλειστές πόρτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεύτερη κέρια εξέλιξη, το ανέφερα και προηγουμένως, η Επιτροπή ε, γίνεται ο Έλληνα και πιο ισχυρό πολιτικό ε, φορέας. Και κάποιε ενδείξει γι' αυτό είναι ότι η Επιτροπή Γιούγκερ αντικατοπτρίζει μια μεγάλη συμμαχία ε, συντηρητικών, σοσιαλδημοκρατών και φιλελευθέρων. Ο Σοσιαλδημοκράτη είναι ο πρώτο αντιπρόεδρο τη Επιτροπή. Εκπροσωπούνται και οι φιλελεύθεροι. Υπάρχει λοιπόν μια ευρεία συμμαχία. Έχουμε κάποιες ομαδοποιήσεις των αντιπροέδρων που είναι άλλο καινοτόμο στοιχείο αυτής της Επιτροπής με πρώην αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στους αντιπροέδρους με ειδικέ αρμοδιότητες. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα λειτουργήσει πρακτικά. Εγώ το στηρίζω, νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε τέτοιε ομαδοποιήσεις. Δεν ξέρουμε όμως αν θα λειτουργήσει καλά. Θα το δούμε στην πράξη. Και αν ε, δεν λειτουργήσει καλά από την αρχή, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ολόκληρο το σύστημα. Και τέλος βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Γιούγκερ θέλει να διαδραματίσει πιο σημαντικό πολιτικό ρόλο. Ακόμα και ενώπιον επιμέρους κρατών μελών. Αν δείτε την ε, ε, έντονη αυτή ρητορική που ακολούθησε τις ιδέες και προτάσεις του, δηλαδή να αξιοποιούνται μέσα από τον ESM για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων επενδυτικών. Αυτό δείχνει ότι θέλει να έχει πιο σημαντικό πολιτικό ρόλο. Και ήδη συμμετέχει ως ε, μελλοντικός πρόεδρος της Επιτροπής στην πολιτική των κρατών μελών. Το έχει κάνει ήδη δύο φορές το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει όμως και μια αντίθετη δύναμη ε, που επιδρά σε αυτή την ε, στρατηγική πόλωση και πολιτικοποίηση. Κάτι το οποίο ε, θεωρήθηκε αρνητική εξέλιξη. Ακούσαμε σημαντικές επικρίσεις και δημόσια και πίσω από κλειστέ πόρτε για την διαδικασία εκλογής ε, του Προέδρου. Πολλοί φοβούνται στα κράτη-μέλη ότι ξεφεύγει από κάθε έλεγχο το σύστημα, ότι κινείται προς μια κατεύθυνση που δεν θα μπορούν πλέον να επηρεάσουν. Και υπάρχει και ο φόβος πολιτικού ευνοχισμού σε πολλά κρατημέλη. Συγγνώμη για την έντονη διατύπωση. Τώρα πώς ε, θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη δεν ξέρουμε. Ενδιαφέρουσα θα είναι η σύνδεση μεταξύ του κυρίου Τούς και του Προέδρου της Επιτροπής, του κυρίου Γιούνκερ. Πώς ε, θα υπάρχει, πόσο, τι μορφή θα πάρει αυτή η επαφή ή η συνεργασία στο μέλλον. Όλα καλά πήγαν με τον κύριο Βαρόσο και τον κύριο Βαν αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά το τζιν έχει βγει από το λιχνάρι. Και όλοι βλέπουμε ότι υπάρχουν και πιθανά αρνητικά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας στο μέλλον. Υπάρχει λοιπόν τέτοια πιθανότητα, αλλά έχει αν έχουν ανοίξει οι ασκοί του αιώλου, δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να τους ξανακλείσουμε. Πρέπει να δούμε προ τα πού θα κινηθούν και να μην νοσταλγούμε το παρελθόν. Κλείνοντα. ας εξετάσουμε τις μελλοντικέ προβλέψεις. Τι μορφή θα μπορούσε να λάβει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό το εγχείρημα, αλλά θα προσπαθήσω. Εντάξει, βέβαια, με κάθε επιφύλαξη, γιατί είναι μεγάλη αβεβαιότητα. Υπάρχει ένα γενικό κλίμα στις Βρυξέλλες ε, και στις πρωτεύουσες των μελών ε, που κινείται με γνώμονα το γεγονός ότι πολλά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ένα κλίμα ότι έχουμε περάσει τα χειρότερα, μια τέτοια ατμόσφαιρα. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό, αλλά γενικά αυτή η αίσθηση υπάρχει. Και ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να ε, πιάσουν τόπο αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει. Και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να τις εφαρμόσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και αν θέλουμε να πάμε ακόμα παραπέρα, το να είμαστε πιο φιλόδοξοι τελικά μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραν. Και ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να κάνουμε κέρια σημασία μεταρρυθμίσει. Γιατί υπάρχει αρνητικό κλίμα σε πολλά κρατημέλη και ότι το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα, στην ανάπτυξη, στην ε, απασχόληση. Το μότο λοιπόν είναι να κάνουμε λιγότερα αλλά καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Και αν δείτε τις προτάσεις επιτάπητος ε, το 2012, το blueprint της Επιτροπής, ε, όλα αυτά τα ζητήματα δεν ε, συζητιούνται καν. Για τις ε, θεσμικές μεταρρυθμίσεις υπάρχουν και εδώ επιπτώσεις, ότι έχουμε λοιπόν ε, αυτό το πνεύμα της μεταρρυθμιστικής κόπωσης εντός οργανικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει όρεξη για νέε μεταρρυθμίσει. Πολύ φοβούνται ότι θα ανοίξουμε το κουτί τη Πανδώρα, ότι θα έχουμε νέε ε, αλλαγές ε, της συνθήκης, ότι θα υπάρχει δυσκολία να καταλήξουμε σε συνένεση μεταξύ των 28 κρατών μελών και φόβοι και ανησυχίε σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε κύρωση στα κρατημέλη, Ήδη είναι νοπέ οι μνήμε από την περασμένη φορά. Τι θα γίνει λοιπόν στα επόμενα χρόνια, μάλλον θα πρέπει ε, να ε, περιοριστούμε και να αρκεστούμε στην σταδιακή αυτή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Άκουσα και διάβασα και τα σχόλια του κυρίου Ντεσκουτέτα και σίγουρα θα αναφερθεί σε αυτά όταν θα αναφερθεί σε συγκεκριμένα ε, παραδείγματα. Αυτά θα έχουμε όμως μικρές αλλαγές εδώ και εκεί, τίποτα το πολύ σημαντικό. Ξεκίνησα περιγράφοντας την κατάσταση σήμερα και τις στρατηγικές προκλήσεις. Εάν ισχύουν όλα αυτά που είπα, ότι ο κατακαιρματισμός και η απώλεια αυτής της αίσθησης ε, της ε, αμοιβαίας ωφέλειας για όλους, αν ισχύουν όλα αυτά λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή να περάσουμε σε πιο ουσιαστικές αλλαγές. Όχι τώρα, αλλά κάποια στιγμή. Τι θα γίνει τότε δεν ξέρω. Υπάρχουν όμως κάποιες ενδείξεις, αν δείτε στην ε, συνθήκη ε, δημοσιονομικής σταθερότητας, βλέπουμε ότι θα πρέπει μέχρι το 2018 να προχωρήσουμε με ουσιαστικά βήματα. Βλέπετε όμως ότι σε κάποιο σημείο χρονικά θα υπάρξει αυτή η αλλαγή στη συνθήκη, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προετοιμασίες για αυτό <clears throat> και αυτό απαιτεί τη δημιουργία μιας καλύτερης ατμόσφαιρας, ενός καλύτερου κλίματος για να δημιουργήσουμε μια νέα συμφωνία, ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της για να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι δεν είναι πια παιχνίδι θετικού αθρίσματος η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να περάσουμε και στην εξέταση των λεπτομεριών για αυτή την αλλαγή, την εντολή και του, τον τρόπο δημιουργίας μιας συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης και να δούμε τι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις θα μπορέσουν να γίνουν. Δεν ξεκινάμε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις που θα θέλαμε, αλλά με τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμόσουμε για να προχωρήσουμε και που δεν μπορούν να γίνουν με την τωρινή συνθήκη. Εδώ θέλω να κλείσω λοιπόν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω λοιπόν ε, αν θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο ε, για τις προκλήσεις, αλλά ήσασταν πολύ ρεαλιστικός. Θα δώσω τώρα το λόγο στον καθηγητή Φαντεσφάν για να λάβει το λόγο και μετά στον κύριο Τισκουτέτε, ο οποίος μόλι ήρθε και τον οποίο χαιρετάμε και καλωσορίζουμε. Ποιο μικρόφωνο να πάρω, λέει ο καθηγήτη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω προετοιμάσει μια πάρα πολύ σύντομη παρουσίαση PowerPoint. Ελπίζω θα είναι αναγνώσιμη στην οθόνη. Εγώ θεώρησα, ερμήνευσα μάλλον διαφορετικά την πρόσκλησή σας από ότι ο προηγούμενος ομιλητής. Είδα και την ημερήσια διαταξή σας και είδα ότι είχατε την επαφή με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών. Γι' αυτό επίτηδες ακολούθησα και την αίτησή σας να εστιάσω περισσότερο στα θεσμικά θέματα, αλλά στα θέματα που δεν απαιτούν αλλαγές ε, στη συνθήκη Γι' αυτό θέλησα να αντιμετωπίσω μια σειρά από θέματα τα οποία είναι ουσιαστικού χαρακτήρα γιατί εσείς εκπροσωπείτε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά επίσης και είσαστε φορείς της νομιμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί υπάρχουν προβλήματα πολλές φορές στην επαφή με τους πολίτες. Ως ακαδημαϊκός λοιπόν θέλω να θέσω όλα αυτά τα θέματα επιτάπητος τα οποία τα γνωρίζετε ενδεχομένω, αλλά για να επιβιώσει το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να φέρουμε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στον απλό πολίτη. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω στα επόμενα 15 λεπτά. Τα τρία θέματα λοιπόν, η νομιμοποίηση, η υποστήριξη της δημοκρατίας και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να διεξέλθω. Και θέλω να πω και ορισμένα θέματα, να θίξω ορισμένα θέματα για την περίπτωση που δεν θα έχουμε να κάνουμε επαναστατικές αλλαγές στην ε, Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι θα μπορούσε να γίνει και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και να σταθώ επίσης και στο θέμα της συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί στη συζήτηση που κάνατε με τον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου, εγώ κατέγραψα το γεγονός ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια για τους δικούς τους θετικούς ε, λόγους έχουν αρχίσει να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην διαδικασία λήψης απόφασης και θα χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία της ε, κίτρινης, πορτοκαλί ή ακόμα και κόκκινης κάρτας που μπορεί να οδηγήσει στην ε, διακοπή των διαπραγματεύσεων για ένα νομοθέτημα. Εγώ θα ήθελα να δω τα Εθνικά Κοινοβούλια από μια διαφορετική οπτική γωνία, την οπτική γωνία της συνεργασίας, όχι της αντιπαράθεσης. Αυτά τα οποία λοιπόν θέλω να σας πω είναι απλά και ταπεινά, αλλά Θέλω να αναφέρω και δύο θέματα, να αναφερθώ σε δύο θέματα που δεν θα γίνουν επίκαιρα στο άμεσο μέλλον, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και εδώ σκέφτομαι συγκεκριμένα την δική σας εμπειρογνωμοσύνη στα συνταγματικά θέματα. Πρέπει λοιπόν να τα αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα και πρόκειται για την συνεργασία και την απλοποίηση των διατάξεων και των προϊόν της και θέλω να μιλήσω εδώ για το θέμα αυτού που ονομάζω διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λόγω του αριθμού των κρατών μελών και των δυσκολιών που αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα και ίσως θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Είμαι οπαδός βέβαια της διεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε τώρα ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών, 28, και είναι πολύ διαφορετικές οι χώρες αυτές στη φύση τους και υπάρχει μια ετερογένεια που θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Και αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει στην, ε, ε, στην παρουσίαση PowerPoint αφορούν μόνο τα δύο τελευταία στοιχεία. Οπότε θα ξαναγυρίσω στο θέμα των εκλογών και το θέμα της νομιμοποίησης, υποστήριξης των πολιτών και της δημοκρατίας γενικά. Η προσέλευση των εκλογέων στις τελευταίες εκλογές ήταν περίπου 42,54%. Ε, Εντάξει, δεν είναι άσχημα, αλλά θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και καλύτερα. Αν λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο που έχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι να έχουμε καλύτερη προσέλευση των εκλογέων. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Και αυτά είναι απλώς ιδέες, οι οποίες δεν απαιτούν κάποια τροποποίηση των συνδικών. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γίνει πιο ορατό στα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Έχετε πολλά καθήκοντα, πολλές ευθύνες, αλλά ένα από τα κύρια θέματα τα και θέματα που θα είναι σημαντικά στο έμεσο μέλλον, στο άμεσο μέλλον και μεταγενέστερο μέλλον, είναι η παρουσία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μονάχα ατομικά στις εκλογικές του περιφέρειες, αλλά και μια πιο διαθρωμένη παρουσία που να γίνεται πιο ορατή για τον απλό πολίτη. Γι' αυτό σας προτείνω να οργανώνετε σε πιο τακτική βάση συναντήσεις εμπειρογνωμών από τη δική σας πλευρά με εμπειρογνώμονες από τα εθνικά κοινοβούλια. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να έχετε συζητήσεις, συναντήσεις, συνδιασκέψεις μέσα στα πλαίσια συναντήσεων πολιτικών ομάδων, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει και μεγαλύτερη ορατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διάφορα κράτη-μέλη οι τακτικές λοιπόν συζητήσεις που οργανώνονται μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια, στα Εθνικά Κοινοβούλια <clears throat> ή με την ευκαιρία δημοσίων ακροάσεων με εμπλεκόμενους παρόντες, αυτό είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμπειρογνώμων σε επίπεδο των επιτροπών, σε επίπεδο πολιτικών ομάδων, στα κοινοβούλια, σε δημόσιε ακροάσεις, να κατεβείτε και στον δρόμο να το πω έτσι και φυσικά τα μέσα ενημέρωση να είναι παρόντα για να μπορέσει αυτή η πληροφορία να φτάσει στην κοινή γνώμη για το θέμα της δημοκρατίας. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη ε, σημασία στο θέμα αυτό των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λέει η συνθήκη ότι συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή συνειδητοποίηση και εκφράζουν την άποψη των πολιτών. Αλλά ξέρουμε όλοι πόσο πολύπλοκο είναι αυτό και ιδίω ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν και τα εθνικά κόμματα για τα θέματα αυτά. Αλλά ίσως η λύση δεν είναι να δημιουργήσουμε αμέσως ευρωπαϊκά κόμματα. Νομίζω στις τελευταίες ευρωεκλογές οι εκστατείες έγιναν και επί τη βάση μανιφέστων, κοινών προγραμμάτων με ένα περιορισμένο αριθμό κοινών σημείων από ευρωπαϊκά κόμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά όμως δεν ήταν ιδιαίτερα ορατά σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο κρατών μελών. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω υπέρ του να κάνουμε σαφείς επιλογές. Εδώ στέκονται οι χριστιανοδημοκράτες, εδώ είναι οι σοσιαλιστές, εδώ είναι οι φιλελεύθεροι και να ζητήσετε από τους εταίρους σε εθνικό επίπεδο, φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές κτλ. να πάρουν αυτά τα προγράμματα, να τα παρουσιάσουν στην εθνική κοινή γνώμη και στις εκλογικές τους περιφέρειες και να τα αναγορεύσουν σε στοιχεία εθνικής συζήτησης όσο προσεγγίζουμε τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουμε όλοι, αλλά είμαι πεπισμένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα και πιο διαρθρωμένα για να επιτύχει μεγαλύτερη ορατότητα και ιδίως εδώ πρέπει να μεταλαμβαδευτούν οι πεπιθήσεις σας και τα προγραμματικά στοιχεία που σας ενδιαφέρουν και φυσικά και τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να βοηθήσουν να φτάσουν οι δικές σας απόψεις στον απλό πολίτη. Αυτό είναι θέμα της ε, δημόσια ευθύνες των μέσων ενημέρωση που είναι γενικά ιδιωτικοί φορείς. Τώρα όταν, όταν ερχόμαστε στι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το άμεσο μέλλον θέλω να αναφέρω μία σειρά από θέματα. Έχετε βέβαια ένα είδος δικαιώματο πρωτοβουλία. Όπω αναφέρεται στο άρθρο 225 τη Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Κομισιόν να υποβάλει μια πρόταση σε θέματα που θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να τύχουν δράσει υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εφαρμογή των συνδικών. Μπορώ να φανταστώ στο μέλλον, λαμβάνοντα υπόψη και την κρίση που έχουμε περάσει και α ελπίσουμε ότι έχουμε φτάσει στο τέλο τη σύραγγο, για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής πολιτικής, εκεί θα μπορούσατε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες και να δείτε σε ποιο βαθμό υπάρχει περιθώριο να διερευνήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το είδος δικαιώματος πρωτοβουλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το ίδιο ισχύει για την απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης των συνδεκών. Και εκεί έχετε το δικαίωμα της πρωτοβουλίας σε σχέση με το άρθρο 48 παράγραφος 7 όταν πρόκειται να υπάρξει ένα τμήμα να υπάρξει μεταρρύθμιση ενός τμήματος των προνοιών του άρθρου 3. Εκεί λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ουσιαστικά το δικαίωμα πρωτοβουλίας για να μπορέσει να επιφέρει <clears throat> τις τροποποιήσεις αυτές οι οποίες είναι προσφυλή στο ίδιο το Κοινοβούλιο. Και ένα δεύτερο στοιχείο θα πρέπει να σας ενδιαφέρει, ότι υπάρχει η αναφορά στην αλλαγή από ομοφωνία σε ειδική πλειοψηφία σε ορισμένου τομεί και επίσης η δυνατότητα, οι εξειδικευμένες διαδικασίες να μεταμορφωθούν στην τακτική νομοθετική διαδικασία και αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει και αν έχετε λοιπόν μια επιστημονική νομοπαρασκευαστική υπηρεσία μπορείτε να συζητάτε μαζί τους και να κάνετε επιλογές για το τι θα κάνετε στα θέματα αυτά τώρα σε σχέση με τις εποπτικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θέλω να επαναλάβω τη συζήτηση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου για το θέμα του ελέγχου της Κομισιόν. Έχετε δυνατότητα να ελέγχετε την Κομισιόν συλλογικά, η οποία είναι υπεύθυνη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει ο πρόεδρος της Επιτροπής μάλλον, μετά από κάθε συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ίσως και το Συμβούλιο μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο στο τομέα του να διαβουλεύετε με το Κοινοβούλιο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Θα πρέπει ο ή η η ειπατη εκπρόσωπος να σας πληροφορεί για όλα αυτά τα θέματα. Τέλος, οι αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με την δυνατότητά σας να πράξετε ως εκλεγμένοι ε, εκπρόσωποι. Και εδώ ως ανεξάρτητος ακαδημαϊκός θέλω να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πείραμα των Spitzenkandidaten. Είναι κάτι που δείχνει το τι μπορεί να πετύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά, σας το λέω πάλι ως απλός πολίτης προσωπικά, με εξέπληξε κάπως ο βαθμός της πολιτικοποίησης που έγινε στις ε, ακροάσεις ορισμένων επιτρόπων. γιατί δεν υπάρχει αυτή η άμεση διαδικασία εκλογής από τους πολίτες για τους επιτρόπους. Επομένως, η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αυτό το καταγράφει η συνθήκη, το Κοινοβούλιο θέλει, πρέπει να δώσει την έγκρισή του στο σύνολο της Επιτροπής, ως συλλογικό σώμα. Ακόμα, για μένα αυτό σημαίνει, ότι ο κάθε υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται ενώπιον σας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε σχέση με την ικανότητά του σε θέματα ουσίας και όχι σε σχέση με την πολιτική προέλευση του κάθε <clears throat> υποψηφίου. Αλλά σε κάποιες ακροάσεις το στοιχείο της πολιτικής προέλευσης έπαιξε κάποιο ρόλο. Πιστεύω, κατά τη δική μου άποψη, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εξετάζει και να διερευνά την εμπειρογνωμοσύνη αυτών των ανθρώπων και όχι τόσο πολύ τις πολιτικές τους απόψεις. Ε, μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω για, τις, ε, για περαιτέρω θέματα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση υπάρχει μια πολύ σημαντική συμφωνία για τη σταθερότητα και τον συντονισμό στον οικονομικό και νομισματικό τομέα τα κράτη-μέλη έχουν πράγματι προσυπογράψει αυτό το σύμφωνο την ε, υποχρέωση συγκεκριμένα να ενσωματώσουν την ουσία αυτής της συμφωνίας στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συνθήκες, μέχρι την παρέλευση πέντε ετών από την θέση εφαρμογής αυτού του συμφώνου για την ε, οικονομική συνεργασία. Αν διαβάσω καλά την ε, διατύπωση του συμφώνου αυτού, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η μεταγραφή του συμφώνου αυτού μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης δεν χρειάζεται <clears throat> κάποια αλλαγή των συνδικών. Εσείς πρέπει να εξασφαλίσετε ότι αυτή η υποχρέωση όμως θα πραγματοποιηθεί. Και μετά για την ε, Οικονομική Ένωση και την Κοινωνική Ένωση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εκεί πρέπει να δώσετε πολύ περισσότερη έμφαση στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στη συνθήκη που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών να συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές. Υπάρχει επίσης και μια αμνία στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε αυτή τη διαδικασία συντονισμού, περιορισμένη μεν, αλλά έχετε την ευθύνη να παρακολουθείτε πως οι ευρείες κατευθυντήρες γραμμές σε σχέση με την εφαρμογή των πολιτικών αυτών κατευθύνσεων εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη στην πράξη. Για το ρόλο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων έχω ήδη πει στην αρχή ότι αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα η μεγαλύτερη ευθύνη των Εθνικών Κοινοβουλίων συνάπτεται με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου περιθμών 2 τον ε, έλεγχο της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Αυτά τα συζητήσατε και δεν πρόκειται να επεκταθώ περαιτέρω. Εδώ η έκκλησή μου είναι βρείτε και τις δυνατότητες να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στα θέματα αυτά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αρχή της έμεσης δημοκρατίας. Οι πολίτες εκλέγουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά και τα Εθνικά και, τα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουν μια μεγαλύτερη συνεργασία γιατί είναι προ το αμοιβαίο συμφέρον περισσότερο από ό,τι συνεργάζονται τώρα. Για τη σχέση με τα κράτη-μέλη και του άλλου θεσμού, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσετε περισσότερο την δυνατότητα να εμπλέκεστε σε συζητήσεις μεταξύ του, της Τρόικας των Προεδριών και της Κομισιόν όταν θεσπίζουν το πρόγραμμά τους για τα τρία εξάμεινα, εκεί να πρέπει να υπάρχει περισσότερη συμμετοχή και εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην χάραξη προτεραιοτήτων και στη διαμόρφωση αυτού του κοινού προγράμματος για τα, για τα τρία αυτά εξάμεινα. Και τώρα τα τελευταία στοιχεία που ήθελα να τονίσω. Υπάρχει το θέμα της διαφοροποίησης σε επίπεδο ολοκλήρωσης. επειδή θέλετε και εσείς να προβληματιζόσετε για αυτά τα συνταγματικά θέματα, πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο της ενισχυμένης συνεργασίας και εδώ θα ήθελα να σκεφτούμε και για το θέμα της απλοποίησης των ε, προνοιών των διατάξεων της συνθήκης. Αυτό το οποίο ήθελα να σας παρουσιάσω είναι ο αριθμός των κρατών μελών και εδώ υποστηρίζω ότι θέλουμε τη διεύρυνση και θέλουμε να έρθουν και άλλα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πολύ μεγάλε <clears throat> οι διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει μεγαλύτερη ετερογένεια παρά ομοιογένεια. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα λοιπόν διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, το ευρώ, το τομέα τη δικαιοσύνη και των εσωτερικών, η εξωτερική πολιτική και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι βάσει των συνθηκών η ενισχυμένη συνεργασία δεν είναι κάτι το κακό. Είναι κάτι που αναφέρεται σαφώς στις συνθήκες ότι η ενισχυμένη συνεργασία θα έχει σαν στόχο να προωθήσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εμβαθύνει και να ενισχύσει την πολιτική, τη διαδικασία ολοκλήρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα όπου μπορούν να υπάρξουν εν καιρό τροποποίηση τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Προφανώς μια πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο για την ενισχυμένη συνεργασία προβλέπει εννέα κράτη-μέλη. Αλλά χρειάζεται και η έγκριση του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία, προτάσει τη Κομισιόν και αφού έχουν λάβει και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να μην μακρηγορώ, η εντύπωσή μου είναι, κοντολογής, ότι εν ώψη των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών Κάποια κρατημέλη δεν είναι έτοιμα να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν έχουν την ικανότητα να ακολουθήσουν την ταχύτητα ε, άλλων χωρών στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Επομένως, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε για τις διαδικασίες της ενισχυμένης συνεργασίας που μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί μόνο σε τρία πάρα πολύ τεχνικά θέματα και κατά την άποψή μου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναδιατυπώσουμε αυτήν την ε, πρόνοια και να τη μετατρέψουμε στο δικαίωμα μιας ουσιαστικής, ενός ουσιαστικού τμήματος των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 45% των κρατών μελών και 50% του πληθυσμού, αλλά όχι να υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα να υπάρξει μια θετική έγκριση από το Συμβούλιο με μορφή ειδική πλειοψηφία. Γιατί όταν δεν μπορεί να υπάρξει ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο υπέρ μια πρόταση Κομισιόν, είναι πολύ απίθανο να θεωρεί κανείς ότι θα μπορούσε να εγκριθεί η ενισχυμένη συνεργασία. Γι' αυτό σας θέτω αυτή την πρόταση να τη σκεφτείτε μέσα στην ομάδα προβληματισμού της ε, Συνταγματικής Επιτροπής και μια άλλη ε, περίπτωση έχει να κάνει με τις μεταρρυθμίσεις στην ε, συνθήκη. Αυτές τις μέρες φαίνεται ότι αυτό είναι ένα ταμπού. Κανένας δεν θέλει να ανοίξει αυτό το θέμα Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική τομή. Λάμβαντε υπόψη ότι ίσως δεν θέλουν όλα τα κράτη-μέλη να υπάρξει μια αλλαγή. Και τα νέα κράτη-μέλη από τα Βαλκάνια, από την Αλβανία, τη Μολδαβία και άλλες χώρες στην, στην Ανατολική Ευρώπη, δεν είναι προφανές ότι όλα αυτά τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν την ταχύτητα ολοκλήρωσης που μπορεί να επιθυμούν τα κράτη που βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό η δυνατότητα να υπάρξει μια συνένεση για τις τροποποιήσεις των συνθηκών... οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για να υπάρξει η αλλαγή των συνθηκών... και να εγκριθεί και να κυρωθεί από τα κρατημέλη, ίσως θα πρέπει και να σκεφτούμε για μια άλλη προσέγγιση. Αυτά τα βλέπετε ήδη στην, ε, στο Διεθνές Δίκαιο για τις ε, συνθήκες, στην συνθήκη της Βιέννης παραδείγματος χάρη. Δεν νομίζω ότι είναι πια δυνατόν ένα κράτος μέλος να περάσει, να καταθέσει μια τροπολογία της συνθήκης η οποία θα εγκριθεί. Κάθε άλλο χρειάζεται να υπάρχει μια ουσιαστική πλειοψηφία, μια, συγγνώμη, ουσιαστική ομάδα κρατών που να υποστηρίζουν μια ε, τροποποίηση και ίσως να είναι λιγότερη από την τωρινή μνήμα που είναι 21 κράτη από 28 λέει 75%. Αυτό θα πρέπει να εξαλειφθεί και θα πρέπει να εξαλειφθεί και η υποχρέωση να υπάρξει εθνική επικύρωση για όλες αυτές τις συμφωνίες. Κάθε κράτος μέλος και αυτό αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 7, κάθε κοινοβούλιο, κάθε εθνικό κοινοβούλιο θα έχει το δικαίωμα να πει όχι, αλλά εκφράζοντας το δικαίωμα ανησυχηρίας δεν θα μπορούν να εμποδίσουν τα άλλα κρεατή τα οποία θέλουν να προχωρήσουν, παραγωγικά τα 21 από τα 28, να προχωρήσουν. Επομένως, διατηρείται την ιδέα ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να δεσμευτεί εναντίον της θέλησής του. Ενώπιον των δυσκολιών όμως που αντιμετωπίζουμε, εγώ θα ήθελα να υπάρξει ένα ξεπέρασμα του δικαιώματος αρνησικυρίας που είναι το ταμπού σε αυτές τις συζητήσεις. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις, πολλές δυσκολίες για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όπως ξέρουμε οι δυσκολίες υπάρχουν για να υπερκεραστούν από την κοινή λογική και αυτό μπορούμε να περιμένουμε από την Συνταγματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα τα αφήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω αμέσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Την προηγούμενη φορά που ήρθα να μιλήσω ήταν ο Τζόρτζο Ναπολιτάνο στη θέση του Προέδρου. Ε, σας εύχομαι κυρία Πρόεδρε ε, μακρά πολιτική εξέλιξη και ε, εξίσου επικοδομητικό έτσι, μέλλον ε, όσο ο πρόεδρος Ναπολιτάνο. Νέες διαπραγματεύσεις για νέα συνθήκη και κατά πόσον αυτό θα ήταν μια ανούσια και ενδεχομένως επικίνδυνη διαδικασία. Νομίζω ότι η κοινή γνώμη δεν είναι έτοιμη ακόμα για να ακούσει για θεσμικές διαπραγματεύσεις και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, έστω και αν αυτό μπορεί να αλλάξει βεβαίως, αργότερα ε, πιστεύω ότι μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει πλέον να ασχοληθούμε με το βάθεμα ε, των συνταγματικών στοιχείων και με την προσπάθεια να τα κάνουμε πιο αποτελεσματικά και πιο ε, αποτελεσματικά και πιο εύκολα στην χρήση τους από την ε, πλευρά της ε, νομιμότητας ε, και της αποτελεσματικότητας θα δούμε τα πράγματα και επίσης θα πω και δύο λόγια όσον αφορά την διαφοροποίηση, πολύ σημαντικό θέμα και θα τελειώσω αναφερόμενος στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που λειτουργεί μάλλον αποτελεσματικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως στην Ευρωκρίση η οποία ε, ήταν κεντρικό ζήτημα των συζητήσεων του, του, του Συμβουλίου. Εκεί ελήφθησαν σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις που είχαν ε, σημαντικές επιπτώσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη, λειτουργώντας συχνά στο borderline ή ακόμα και εκτός ε, αυτής της borderline των αρμοδιοτήτων ε, των ε, συνθήκων. Πιστεύω ότι ο Χέρμαν Βαν Ρόμποϊ έχει καθορίσει τον ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της Προεδρίας έκανε πολλές ε, συζητήσεις, ε, ε, ήλεγξε την προπαρασκευαστική εργαλεία μέσω διαφόρων διάβλων, π.χ. Σέρπας και προσωπικούς συμβούλους. Επίσης έφτασε σε έξι συμβιβαστικές λύσεις και επίσης ήλεγξε την ε, υλοποίηση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί. Και φυσικά ε, μεγάλωσε, αύξησε την ορατότητα στα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύω ότι αυτό το πλαίσιο ε, το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οδηγεί σε ένα λογικό συμπέρασμα ότι ο ε, διάδοχός του θα ακολουθήσει περίπου την ίδια γραμμή. Όσον αφορά την νομιμότητα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ταυτόχρονα το σημείο συνάντησης των εθνικών ηγετών, αλλά και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το αναφέρει ο Μίλας στο εξαιρετικό βιβλίο του ε, «Passage to Europe» τα κράτη-μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, λογοδοτούν ε, στα κοινοβούλια και στον λαό τους ε, σύμφωνα με τις θεσμικές συμφωνίες. Επίσης γνωρίζουμε από τις συνθήκες ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει την ίδια νομική δικαιοδοσία, συγγνώμη, δο, λογοδοσία απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να καλυφθεί επομένως αυτό το ε, δημοκρατικό έλλειμμα μέσω πιο θεσμοθετημένων και πιο συχνών επαφών. Δεν είναι το ίδιο ε, με την λογοδοσία. Εγώ αναφέρομαι ε, σε πιο σαφείς επαφές και σχέσεις ανάμεσα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, σημείο στο οποίο θα επανέλθω αργότερα. Δύο λόγια όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κανείς δεν αμφισβητεί την ε, ε, νομιμότητα του μόνου άμεσα εκλεγμένου πολυ, ε, πολυεθνικού οργάνου. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό έχει νομιμοποίηση φυσικά. Αλλά θα πρέπει να σχολιάσω τα εξή. Η πυρηνική εργασία ε, κάθε κοινοβουλίου είναι, καθορίζεται από την εκτελεστική ε, εξουσία. Υπάρχει μακρά παράδοση έγκρισης ψηφισμάτων ε, για σημεία που αφορούν το σύνολο των πολιτών. Εγώ θα έκανα μια οικονομική ε, πρόταση ή συμβουλή ε, ορθώς ή εσφαλμένα. Υπάρχει αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο σύνολό τους και γενικά προσπαθούν να ε, διευρύνουν το ε, δικό τους ε, πλαίσιο εργασίας και επιρροής, αυτό που αναφέρεται στον βρετανικό τύπο ως middling. Αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο αναφέρεται στην κρίση και θα το γνωρίζει βεβαίως ο παρακαθήμινος πρόεδρος. Έχει αποδειχθεί ότι πολλές αποφάσεις ε, πρέπει να παίρνονται σε ένα επίπεδο, ενωσιακό ας πούμε ή σε επίπεδο ευρωζώνης, αλλά υλοποιούνται σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο των κρατών μελών. Αυτές οι αποφάσεις συχνά αφορούν οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές ε, πολιτικές οι οποίες είναι ιδιαιτέρως προσφυλείς και βρίσκονται στο κέντρο ε, των τοπικών εθνικών ε, πολιτικών συζητήσεων και επομένως εδώ χρειάζεται δημοκρατική νομιμοποίηση και στα δύο επίπεδα και αυτό θα πρέπει να σημάνει περισσότερο συντονισμό και διάλογο ανάμεσα στην Ευρώπη και τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα ε, συμφωνήσω με τον καθηγητή Οσουάν ότι ένα σημείο το οποίο αφορά τις προσπάθειες που έχουν γίνει ε, ε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ιδιαίτερα πιστικές οι προσπάθειες αυτές, θα πρέπει να φανταστούμε μερικές νέες εφάνταστες λύσεις και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και κάτι, κάτι τέτοιο, μια τέτοια λύση μπορεί να προέλθει μονάχα από το δικό σας ε, θεσμικό ε, όργανο. Και βεβαίως αυτό παραπέμπει και στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Για την Κομισιόν θα είμαι σύντομος γιατί η βασική σκέψη ε, που ακούσαμε προηγουμένως είναι ότι η Κομισιόν ε, ε, είναι υπεύθυνη λογοδοσίας στο Κοινοβούλιο για, όσον αφορά την εσωτερική εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι γνωρίζουμε όλοι και σίγουρα εγώ είμαι προσωπικά πεπισμένος, η Κομισιόν ως έχει είναι πολύ μεγάλη για να μπορεί να λειτουργήσει σαν κολέγιο. Γνωρίζω βεβαίως ότι ε, πρέπει κατά αυτή την έννοια να γίνουν ε, σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες, αλλά θα πρέπει να προηγηθούν θεμελιώδεις αλλαγές στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δουλέψουμε με αυτήν την Κομισιόν, έστω και αν είναι πολύ μεγάλη για να λειτουργεί καλά πρόεδρος ε, Γιούγκερ, ε, ε, και το ανέφερε και ο πρόεδρος Εμμανουηλίδης αυτό, ο πρόεδρος Γιούγκερ λοιπόν αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα εργασίας βάσει clusters έτσι ώστε να μετριαστεί αυτό το εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος. Πιστεύω ότι η πρόταση είναι πολύ καλή. Βεβαίω, η ανθρώπινη φύση είναι αυτή που είναι και επομένως κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το σύστημα ε, θα ε, εφαρμοστεί εύκολα ε, γιατί οι προσωπικοί εγωισμοί είναι πολύ και σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επομένως καταλαβαίνουμε ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Ε, ωστόσο πιστεύω ότι οι πραγματικές προσπάθειες θα πρέπει ε, να καταβληθούν έτσι ώστε κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πιέσει με όλη του την επιρροή έτσι ώστε να στηρίξει σε αυτή τη διαδικασία τον πρόεδρο Γιούνκερ. Δεύτερο, πιστεύω ότι το μέγεθος της Κομισιόν είναι τέτοιο που θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ψήφου. Ε, ε, πιστεύω ότι αυτό το σύστημα της ε, ομοφωνίας, αυτό το σύστημα της συνένεσης παραλύει τις διαδικασίες. Ε, δεν έχει λειτουργήσει τα τελευταία δέκα χρόνια το σύστημα της ε, απλής ε, πλειοψηφίας γιατί λαμβάνοντας υπόψη τις ανισότητες, την ανισομερή σύνθεση της Κομισιόν δεν έχει λειτουργήσει, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει το σύστημα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η Κομισιόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προτείνει το, το, η Κομισιόν να αποφασίσει έστω ανεπίσημα ότι οι προτάσεις που στηρίζονται από μεγάλη πλειοψηφία και τι είναι το τι ε, ε, ονομάζουμε μεγάλη πλειοψηφία large majority αυτό θα πρέπει ε, να το αποφασίσουμε. Αυτό το οποίο λοιπόν προτείνει η μεγάλη πλειοψηφία θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Αυτό μπορεί να αποφασιστεί εσωτερικά από την Κομισιόν. Και νομίζω ότι ε, το, ε, η εγγενής δυνατότητα βέτο στην παρούσα ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται εν μέρη στη βάση της της ε, κακής ας πούμε επίδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια σε πολλά θέματα. Το τελευταίο που έχω να πω για την Κομισιόν είναι ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο παρούσα στις εθνικές πρωτεύουσες. Οι σημαντικές αποφάσεις δεν θα πρέπει απλά να ανακοινώνονται από έναν ε, ε, απλό εκπρόσωπο της Κομισιόν ε, πίσω στην αίθουσα τύπου ας πούμε της Κομισιόν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παρουσιάζεται από τα ίδια τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις, στις αρμόδιες επιτροπές, στα αρμόδια φόρα και ενώπιον του τύπου από τους ίδιους τους επιτρόπους. Είναι δύσκολος στόχος, τον οποίο όμως πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να τον επιδιώξουμε, γιατί έτσι θα γίνουν πιο κοντινές και λιγότερο, και λιγότερο αναμειγνυόμενες στα εσωτερικά της χώρας αυτές οι αποφάσεις. Θα, θα γίνουν λοιπόν πιο εύκολα αποδεκτές ενδεχομένως. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση τώρα με διάφορα ονόματα και διάφορες ε, απόψεις ε, που ε, ανέρχονται στις διάφορες μορφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μπενελούξ, Σέγγεν, ε, εκεί προβλέπονται διάφορες μορφές, ε, συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία έκανε μια μεγάλη, ένα μεγάλο και διαφορετικό ε, βήμα προς την νομισματική ένωση, οδηγώντας τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο opt-out σε σχέση με την κοινώς αποδεκτή νομική μορφή, συγγνώμη, νομισματική μορφή που θα είχε η Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οδηγηθήκαμε σε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων που λαμβάνοντας υπόψη την στιγμή, τον τρόπο, τον επίπεδο έχει διαμορφώσει ένα ε, πολυεπίπεδο ε, σύστημα ε, στα πλαίσια του οποίου δεν είναι ταυτόσιμες οι απόψεις τις οποίες μοιράζονται όλοι. Βεβαίω, η πολιτική πραγματικότητα είναι αυτή που είναι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκύπτει βεβαίως και από τις ε, ε, διαδικασίες πολλών διευρύνσεων. Εν πάση περιπτώσει, πολλές μέθοδοι θεωρούνται μη ορθόδοξες και ε, σε μερικές περιπτώσεις ότι παραβαίνουν σοβαρά τον κανόνα. Ε, εγώ ε, ε, θα ήθελα να πω ότι αυτού του είδους οι παραβιάσεις εννοούνται λίγο με τον τρόπο που το σεξ εννοείται στην Βικτοριανή Αγγλία. Δηλαδή ξέρουμε υπάρχει, το έχουμε, το κάνουμε, αλλά παραμένει ε, παραμένει στα πλαίσια μίας ασαφούς διατύπωσης. Δηλαδή το κάνουμε αλλά δεν το λέμε, δεν το λέμε με το όνομά του. Και εν πάση περιπτώσει έφτασε η ώρα ε, να γίνει το coming out, να μιλήσουμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνει και γιατί είναι χρήσιμο έτσι ώστε να ε, υπάρξει μία ε, ε, διαφοροποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόνο δύναμη μπορεί να δώσει. Σε σχέση με αυτό που είπε ο πρόεδρος Βαν Ρόμπο, ότι η Ευρώπη έχει δύο καρδιές, το, την ενιαία αγορά και το ενιαίο νόμισμα. Είναι ε, η καρδιά είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Τώρα το να έχεις ε, δύο καρδιές ε, δεν ξέρω εάν είναι καλό ή λάθος. Αυτό παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Αλλά βεβαίως οι δύο καρδιές είναι διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αφενός δεν πρέπει να λησμονούμε και αφετέρου είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει θεσμικές συνέπειες οι οποίες εν λαμβάνονται υπόψη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί τώρα υπάρχουν ε, ε, οι διασκέψεις κορυφής. Θυμάμαι ότι το 2008 αυτό ε, θεωρήθηκε απολύτως ανορθόδοξο και απαράδεκτο, ενώ τώρα είναι, είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινή ζωή, αυτές οι διασκέψεις της Ευρωζώνης. Είναι μια ε, ζώνη, οποία, ευρωζώνη η οποία έχει και το δικό της ε, πρόεδρο ε, και επομένως βλέπουμε ότι έχουν προσαρμοστεί όλοι σε αυτήν την διαφοροποιημένη κατάσταση. Μέχρι έναν βαθμό πιστεύω ότι η Κομισιόν μέσω του, του, συλλογικού χαρακτήρα της προσπαθεί να βρει λύση σε αυτό το διαφοροποιημένο περιβάλλον και εκπλήσωμε ε, βέβαια που ο πρόεδρος της Ευρωζώνης πλέον ε, ε, είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από μια χώρα που δεν συμμετέχει στην Ευρωζώνη γιατί θα αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα επόμενη ας πούμε καμπή της διαφοροποίησης. Επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς και με ποιο τρόπο θα, επηρεαστεί η πραγματική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα αυτά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαβουλευθεί επί νομικών πράξεων και πολιτικών που επηρεάζουν μόνο την Ευρωζώνη. Το Κοινοβούλιο ισχυρίζεται ότι δικαιούται να παρεμβαίνει σε αυτά τα ζητήματα ως ε, νόμιμος και δημοκρατικός εκπρόσωπος ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται για μία θεραλέα διατύπωση και δήλωση, κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι θα αμφισβητηθεί κάποιες φορές αυτή η δήλωση. Το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει την εσωτερική του οργάνωση ε, σε μια ισχυρότερη, πολυεπίπεδη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και καλό θα ήταν να το εξετάσετε. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα δεν θα επιληθεί αν το αγνοήσουμε. Κλείνοντας, για την εμπιστοσύνη. Εκπλήσωμε με το επίπεδο με, το έλλειμμα εμπιστοσύνης με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι σήμερα. Μιλώ για έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ εθνικών και ενωσιακών θεσμικών οργάνων. Έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και έλλειμμα εμπιστοσύνης βεβαίως μεταξύ κρατών μελών μεταξύ των, ε, των ins και των outs, των μέσα και των έξω και η εμπιστοσύνη για τη δυνατότητα ε, εφαρμογής υλοποίησης του ευρωπαϊκού οράματος ε, είναι ελλειπής και βεβαίως έχουμε χάσει και την αυτοπεποίθησή μας. Αυτό το ζήτημα λοιπόν της εμπιστοσύνης και της αυτοπεποίθησης, έδωσα και μερικά παραδείγματα μόλις τώρα, θεωρώ ότι λειτουργεί ως τροχοπέδι ε, ως προς την ε, εύρυθμη λειτουργία των ε, θεσμικών οργάνων και αποτελεί κίνδυνο. Αυτά τα επίπεδα έλλειψης εμπιστοσύνη συνιστούν κίνδυνο για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Και νομίζω ότι αυτό το θεσμικό όργανο είναι σε καλύτερη θέση από οποιοδήποτε άλλο να κάνει κάτι για αυτό το ζήτημα. Να εξετάσει, να αναλογιστεί πώς μπορεί να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ίσως πρέπει να συναγάγουμε συμπεράσματα από αυτή την υπόθεση, να εξετάσουμε ε, αυτό που υπόθηκε για τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί έτσι μπορεί να μειωθεί ε, η δυσπιστία μεταξύ των ε, θεσμικών αυτών οργάνων. Πρέπει να αποτελέσει ε, κύρια προτεραιότητα, ειδικά για τον Νότο. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Ε, είχαμε τρεις εξαιρετικές και πολύ καλά τεκμηριωμένες ε, εισηγήσει. Ξέρω ότι έχει περάσει η ώρα, αλλά να δώσουμε το λόγο στα μέλη μας. Ο κύριος Σέπφλιν έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους τρεις ε, ομιλητές. Θα ήθελα να επανέλθω αρχικά στα όσα είπε ο κ. Μανουλίδης. σε ένα βαθμό θεωρώ ότι αυτό ισχύει και για τις τρεις ε, παρεμβάσεις. Το ζήτημα της εμπιστοσύνη. είναι μία από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Ιδίως οι ανισότητες που εντείνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, αφορούν το καθεστώς, την πρόσβαση στην εξουσία και ούτω καθεξής. Και εδώ θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που ανέφερε ο κύριος Πρέσβης. Η εμπιστοσύνη αντικατοπτρίζει εν μέρη την θεσμική ισχύ και τη διαφάνεια. Και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε έλλειψη αυτής της εμπιστοσύνης. Γιατί ο κόσμος δεν δέχεται ότι ε, οι, τα θεσμικά αυτά όργανα λειτουργούν προς όφελός τους, προς το συμφέρον τους. Είναι μακριά δεν έχουν πρόσβαση είναι αδιαφανή. Και υπάρχει και αυτή η ορολογία, αυτές οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ουσιαστικά δεν μεταφέρουν το μήνυμα ε, στο ευρύ κοινό. Αυτά που αποδόθηκαν προηγουμένω για την μεγαλύτερη προβολή ε, στα κράτη-μέλη. Πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά η εμπειρία μου στην Ουγγαρία δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Τα μέσα μαζική ενημέρωση ενημέρωση στα οποία αναφερθήκατε, απλώς δεν δέχονται ότι ασκείται ε, πραγματική εξουσία στις Βρυξέλλες. Δέκα χρόνια σε αυτά τα θεσμικά όργανα με έχουν πείσει ότι είναι απίθανο να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Και πάλι, εν μέρει αυτό ε, οφείλεται στην ε, ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, αλλά και στην πολύπλοκη αυτή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Είναι σχεδόν απίθανο, θεωρώ, να περάσουμε από αυτόν τον σχετικά μικρό κύκλο εμπειρογνώμων που κατανοούν την οικονομική διακυβέρνηση. Όσοι δεν την κατανοούν, δεν μπορούν να ε, την εμπιστευθούν. Δύο ερωτήματα. Γιάννη, μίλησες για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι πλέον σε θέση να εξισορροπήσει τα εθνικά συμφέροντα. Νομίζω ότι σωστά παρέθεσα τα όσα είπες. Κατά τη γνώμη σου, πώς συνδέεται αυτό με την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μηχανισμός επίλυσης διαφορών, που είναι κύρια αρμοδιότητα και λειτουργία από την ίδρυσή της Ένωσης. Επίσης, μίλησατε για το νέο πρότυπο, το νέο φυσιολογικό. Τι εννοείται με πολιτικοποίηση και τι είδους πολιτικοποίηση εδώ, εννοούμε εδώ. Δεν ε, το ε, ξεκαθαρίσατε, χρησιμοποιήσατε αυτόν τον όρο, αλλά ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε με αυτόν τον όρο. Και σε ό,τι αφορά αυτό το, την, το νέο κλίμα ε, των σταδιακών αλλαγών, σίγουρα θα γνωρίζετε το επιχείρημα Φουκουγιάμα για την... Ε, ε, πολιτική αποσάθρωση ε, και παρακμή. Αυτό συμβαίνει όταν τα θεσμικά όργανα δεν ανταποκρίνονται πλέον στις κοινωνικές αλλαγές, πολιτικές φιλοδοξίες και την αποσύνδεση. Και απόδειξη εδώ είναι οι τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές. Και έχουμε και την αύξηση διαφόρων τάσεων αντιευρωπαϊκών στα κράτη-μέλη. Πολλά ερωτήματα λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουδάντοφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Έχω και εγώ να κάνω ένα σχόλιο καθώς και μία ερώτηση, αλλά έχω και μία πρόταση. Και οι τρεις ομιλητές αναφέρθηκαν σε αυτά που είπε ο πρώτος ε, ε, ομιλητής. Μίλησε για την περιφέρεια της Ευρώπης και την επίπτωση των κρίσεων. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Γαλλία είναι περιφέρεια στην Ευρώπη. Αν δείτε αυτούς που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο φόβος τόσο ευρέως ώστε να υπονομεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματική πηγή της κρίσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστάθειες, είναι η κρίση του κράτους ευμάρειας τα πιο πλούσια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν και το αίτιο της κρίσης του 2012 και οδήγησε στην κρίση σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Η κρίση φαίνεται να προέρχεται από τα πλουσιότερα κράτη. Δεν ήρθε από τα κράτη-μέλη που είναι στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> για τη νέα μορφή τώρα που παίρνει η Κομισιόν υπό τον κύριο Γιούνκερ, το αν αυτό το σχήμα θα αποδειχθεί ισχυρότερο ή όχι. Βέβαια, Έχουμε την προσωπικότητα του κυρίου Γιούνκερ στην Προεδρία της Κομισιόν και τον κύριο Τάσκ, ο οποίος προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα πρέπει να συνεργαστούν. Θα πρέπει να δούμε τώρα το στοιχείο της συλλογικότητας στη συνεργασία τους. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει κάποιος τρόπος με τον οποίο η Κομισιό θα μπορούσε να συνεργαστεί καλύτερα με τα άλλα θεσμικά όργανα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να διοργανώνουν συζητήσεις στα εθνικά κράτη. Γιατί στα εθνικά κράτη οι συζητήσεις αφορούν τα εθνικά πολιτικά θέματα και είναι αντιπαραθέσεις των εθνικών πολιτικών κομμάτων και για την αλλαγή των συνδικών τι θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει αλλαγές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι λιγότερο διάφανο στη δράση του από πολλά εθνικά κοινοβούλια. Και εμεί είδαμε πρόσφατα τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο διορισμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αυτό δεν ήταν μια πολύ σαφής διαδικασία και δεν ξέρω αν και η επιλογή του κ. Γιούνκερ ήταν απόλυτα διάφανη θα πρέπει εμείς να λογοδοτούμε στους πολίτες μας και ξέρουμε πολλές φορές ότι μερικοί από τους στόχους που τίθενται δεν θα επιτευχθούν. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο διάφανοι. Ευχαριστώ. Ο Γιολάινεν. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές ε, για, την, ε, για τις ιδέες που μας έδωσαν. Δυστυχώς έχασα ένα κομμάτι γιατί έπρεπε να πάω στις ακροάσεις. Εμείς θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως ελέγχθη, οι Spitzenkandidaten υπήρξαν εμβληματικές φιγούρες οι οποίες μας προχώρησαν λίγο περισσότερο. Το θέμα είναι τι θα γίνει το 2019. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν ήταν μοναδικό το γεγονός. Το 2014 θα συνεχίσει και στο μέλλον. Εγώ έχω τις δικές μου ιδέες για το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε μια, εθνική, μια ευρωπαϊκή εκλογή, έχουμε 28 εθνικές εκλογές. Και δίκαιο ο Κάμερο που είπε ποιος ήταν ο σπίτσα καντιδάς στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι σωστό. Όταν κάναμε την ε, ε συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, είχαμε μιλήσει για ένα νομοθετικό σύμφωνο, ότι θα μπορούσε ίσως και το Συμβούλιο να αλλάξει τη μορφή του χωρίς αλλαγή των συνδικών και να έχει μια καλύτερη ε, μορφή συντονισμού ανάμεσα στους 16 σχηματισμούς του Συμβουλίου. Και επίσης, προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει θετικό κλίμα για αλλαγές των συνδικών, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μία συλλογική συζήτηση, γιατί τώρα γίνονται εθνικοί εθνικές συζητήσεις, κατακαιρματισμένες συζητήσεις, αλλά τίποτα το συνολικό. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει κάποιο φόρουμ για να συζητήσουμε συνολικά το μέλλον της Ευρώπης και να δούμε τι συμπεράσματα θα μπορέσουμε να αντλήσουμε από αυτό για μια νέα συνθήκη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αρνητικό το ότι δεν έχουμε μια συλλογική συζήτηση. Επίσης, η κρίση μας οδήγησε σε μια εσωστρέφεια. Και αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια πρόκληση. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την θητεία όταν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι πιέσει εκ των έξω προς την Ευρώπη και εμείς παραμένουμε σε αυτήν την εσωστρέφεια. Ο κ. Κατρούγκαλος. Thank Σας ευχαριστώ όλους για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η ιδέα του κυρίου Εμμανουηλίδη για την ε, ασταθή διακυβερνητικότητα σε σχέση με τους θεσμούς. Με τον τρόπο αυτό αντανακλάται ο νέος ρόλος της Γερμανίας σε αυτή την ε, δομή και το δημοκρατικό έλλειμμα που απορρέει από αυτό. Θυμάστε ότι η καγκελάριος ε, Μέρκελ στο παρελθόν καμιά φορά με τον ε, πρόεδρο Σαρκοζή, ανακοίνωνε τις αποφάσεις οι οποίες θα λαμβανόταν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης μέρας. Αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς σοβαρές συνέπειες για τη δημοκρατική νομοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> θα ήθελα όμως σχετικά να ρωτήσω τον καθηγητή Ντεσουάν αν η πρότασή του για μια διεύρυνση της ενισχυμένης συνεργασίας ή του κ. Δισκουτάρη η πρόταση για μια περαιτέρω διαφοροποίηση στη συνεργασία, αν αυτά θα όξυναν περισσότερο την κατάσταση αυτή, δημιουργώντας μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων και έτσι υποσκάπτοντας τη συνοχή και όχι μόνο τη συνοχή, αλλά φυσικά και την πολιτική νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Εμμανουηλίδη για τον ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτό το νέο πλαίσιο που παρουσίασε. Θα ξέρετε ότι ο Επίτροπος Κατάινεν είπε πρόσφατα ότι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν εφαρμόζεται στις χώρες που είναι σε προγράμματα προσαρμογής και λιτότητας με την εποπτεία της Τρόικα. Γιατί κατά την άποψή του τα μνημόνια αυτά δεν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο. Επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα μνημόνια αυτά η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εμένα με εντυπωσίασε αυτή η δήλωση. Γιατί από τη στιγμή που ο χάρτης, η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων βρίσκεται σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου με τη συνθήκη Λισαβόνα, θα περίμενε κανείς το αντίθετο. Και βλέπουμε τώρα να μπαίνουν τελείω σε περιθώριο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα και συγκεκριμένα και η χάρτα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η, ε, ουσιαστικά η θέση στο περιθώριο της χάρτας είναι κάτι το ουσιαστικό γιατί αλλιώς θα είναι κάτι το πραγματικά τρομακτικό. Κύριο Σάντερς. Ένα ερώτημα στον κύριο Ντεσουάν. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα την ε, πρόταση αυτή που είχατε αναφέρει ότι μπορούν να τροποποιηθούν <clears throat> οι συνθήκες χωρίς όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνούν. Να υπάρξουν λοιπόν αλλαγές των συνδικών, αλλά δεν θα ισχύουν στις χώρες αυτές που έχουν ασκήσει το δικαίωμα του βέτο. Μ' αρέσει η ευκαμψία και η μεταβλητή γεωμετρία, αλλά αν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ορισμένα κρατημέλη έχουν ε, δεχθεί τη συνθήκη του Μάστριχτ, άλλα τη συνθήκη της Νίκαιας, άλλα τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και κάποιος συμμετέχει μόνο στην ενιαία πράξη, παραγωγή χάρη, τότε είναι υπερβολικά μεταβλητή γεωμετρία. Είναι πάρα πολλές πρόνοιες στις συνθήκες που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν με μεταβλητό τρόπο και που απαιτούν μια στάθμιση ψήφων στο Συμβουλίο. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να επιληθεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Η Μερσέδες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση και μετά μια σκέψη όσον αφορά την πολιτική διάσταση. Η ερώτηση προς τον Βαρόνο Ντεσούτ είναι γεγονός ότι και το Κοινοβούλιο μπορεί να οργανωθεί ε, επί τη βάση μεταβλητών διαστάσεων. Αλλά μια και το Κοινοβούλιο εκλέγεται άμεσα και μια, σαφώς, μια και σαφώς έχει ενταχθεί κάτι το οποίο ίσως δεν έχει γίνει ακόμα αρκετά κατανοητό και σαφές σε όλους, αλλά εμείς δεν εκπροσωπούμε το κράτος μας, αλλά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό θα ε, δυσκόλευε πολύ την κατάσταση, θα την περιέπλεκε, γιατί η εκλογή κάθε ε, βουλευτή γίνεται επί τη αρχή ε, μιας γενικής εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της χώρας του. Επομένως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα άλλο υποσύστημα, ας πούμε, που θα αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δεν θα αφορά μονάχα μία, ε, μία ομάδα χωρών, ε, γιατί μετά θα έπρεπε να γίνει μία διαφορετική εκλογική αναμέτρηση για τις υπόλοιπες χώρες και θα ήταν πολύ περίπλοκο. Αυτό από πολιτικής απόψεως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Κοινοβούλιο στο ευρωπαϊκό ε, σύστημα. Ε, επί του οποίου σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι, αλλά δυσκολεύομαι να απαντήσω. Δεύτερον, το δεύτερο σημείο αφορά τις ε, ε, διαφοροποιήσεις οι οποίες έχουν που προκύπτουν από την τροποποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας που οδήγησαν σε κάποιες χώρες ε, να και κάποιους υποψήφιους οδήγησαν σε πολιτικοποίηση της ε, ε, εκστρατείας που δεν έγινε απαραίτητα αντιληπτή άμεσα από τους πολίτες αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε αν αυτή η καινοτομία προκαλέσει τροποποιήσεις και στην ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί και την επόμενη φορά ε, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά γιατί ε, σημαντικοί ηγέτες θα μπορούσαν να περνούν από συγκεκριμένες διαδικασίες ας πούμε έτσι ώστε να γίνουν υπεύθυνοι του κόμματός τους μέσα από μια διαδικασία η οποία θα είναι και πιο συμμετοχική και πιο πλήρης σε επίπεδο κρατών. Ωστόσο, το ερώτημα είναι το εξή. Σε ποια τροποποίηση, τουλάχιστον στο ιστορικό των συνθήκων ή ενδεχομένως ε, και μέσα στα πλαίσια μιας νέας συνθήκης, ε, ποιες αλλαγές θα πρέπει να ε, υπάρξουν αυτή η νέα η νέα αρχή εκλογής τουλάχιστον του Προέδρου της Κομισιόν ε, θα αφορά και τη σύνθεση της Επιτροπής, αλλά ίσως θα πρέπει να αφορά ε, και την εντολή της Επιτροπής που θα πρέπει να διαφοροποιηθεί. Επίσης αυτή η πολιτικοποίηση που θα ισχύσει, γιατί κοιτάξτε, ε, προερχόμαστε από από μια περίοδο που η Ευρώπη ειδώθηκε περισσότερο σαν γραφειοκρατία. Αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι πλέον. Ήδη σήμερα η καταγγελίες ε, που γίνονται σε σχέση με την ε, Ευρώπη δεν είναι πλέον γραφειοκρατικού αλλά πολιτικού χαρακτήρα. Κατηγορείται δηλαδή ότι δεν κατάφερε να δώσει λύση στην κρίση. Κοιτάξτε τώρα, τους πολίτες ε, δεν τους ενδιαφέρει πολύ και πολύ λίγα καταλαβαίνουν από, όλα αυτά τα, ε, από όλες αυτές τις ε, συνταγματικές ας πούμε, συζητήσεις. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι δεν κατάφερε να δώσει πολιτικές απαντήσεις στα προβλήματά τους η Ευρώπη. Επίσης, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε περισσότερες εξουσίες μέσα στα πλαίσια των υφισταμένων συνθήκων μπορούμε να βρούμε τέτοιες απαντήσεις στις υφισάμενες συνθήκες, ε, απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών. Διαφορετικά θα πρέπει να βρούμε λύση με ε, άλλο τρόπο. Κατά την άποψή μου, Ήδη ξεπεράσαμε, χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε ξεπεράσει, λέω, την εποχή της γραφειοκρατικής Ευρώπης. Πλέον, η κριτική των πολιτών απέναντι στην Ευρώπη δεν αφορά τη γραφειοκρατία, αλλά την ίδια την πολιτική. Και δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή η κριτική των ε, πολιτών με τις ε, παρούσες δομές και με το Συμβούλιο που έχει όλη την εξουσία από τη μία, αλλά που δεν έχει όμως βάσει του θεσμικού συστήματος άλλες εξουσίες αλλά ούτε και αρμοδιότητες έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει πραγματικές απαντήσεις. Γιατί το διακυβερνητικό μοντέλο δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να διαχειριστεί πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτό είναι ο κόμπο. γιατί στην καθημερινότητα δεν γίνεται αντιληπτή η Ευρώπη ως, μια γραφειο, ε, ως ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, αλλά ως ένας μηχανισμός ο οποίος είναι γραφειοκρατικός και δεν δίνει και πολιτικές απαντήσεις στους προβληματισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και παρεμβάσεις που ακούσαμε. Και νομίζω ότι τις διατρέχει ένας κοινό άξονας που είναι ότι ενδεχομένως δεν είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μεταρρύθμιση των συνδικών. Εν καιρό μπορεί να είναι επιθυμητό κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι από όλε τι παρεμβάσει έχω πάρει το μήνυμα ότι υπάρχουν πολιτικές δυσκολίε και ελοχεύονται κίνδυνοι εάν υπάρξει μια μεταρρύθμιση των συνδικών. Αυτό με οδηγεί στη σκέψη ότι η συζήτηση θα έπρεπε να εστιάσει περισσότερο σε βελτιώσεις στα μικρά ψεγάδια που υπάρχουν τώρα στη συνθήκη. Και το ερώτημά μου είναι, οι μικρές αυτές αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο, κατά πόσο θα επαρκέσουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχουμε ενώπιόν μας, που είναι από τη μία μεριά το πρόβλημα της υπέρβασης της κρίσης και δεύτερον το πρόβλημα του να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη που είναι και η βάση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά συνδέονται με την ε, ανάγνωση που πρέπει να έχουμε των θεσμικών αλλαγών και εξελίξεων τα τελευταία χρόνια. Φοβάμαι ότι αν δούμε ποιες ήταν αυτές οι θεσμικές αλλαγές των τελευταίων ετών και πούμε ότι η κατάσταση κρίσης έχει βελτιώσει την κατάσταση, εδώ πρέπει να πούμε κάτι και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί αλλιώς μπορούμε να κάνουμε ένα σφάλμα, εάν φανταστούμε ότι πέρα από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου που έκαναν πάρα πολλές ώρες και πέρα από αυτές υπήρξε κάποιος άλλος ο οποίος βοήθησε να επιληθεί η κρίση, κάνουμε λάθος. Το γεγονός ότι παρεμβαίνει τώρα η Κεντρική Τράπεζα δείχνει ότι δεν υπήρξε ικανότητα του Συμβουλίου να ξεπεράσει την κρίση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένο δημοκρατικό έλλειμμα. Βλέπαμε κάθε εβδομάδα τον κύριο Ντράγκη να μιλάει στην τηλεόραση και αναρωτιόταν οι πολίτε, τι δημοκρατικό αξίωμα έχει αυτός ο κύριο για να μπορέσει να χαράξει πολιτική. Και γι' αυτό επανέρχομαι στο ερώτημά μου. Ποιες είναι οι θεσμικέ εξελίξεις, οι δυνητικέ θεσμικέ εξελίξεις που δεν αφορούν μονάχα μικρές βελτιώσεις αλλά μπορούν να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε το πρόβλημα της κρίσης και της ανάκτησης της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τέσσερα λεπτά για τον καθένα σας να απαντήσετε. Πέντε λεπτά, αν μας συγχωρήσουν οι διερμηνείς. Αλλά θα αποφασίσετε εσείς ποιος θα λάβει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να απαντήσουμε τόσο πολύ με ερωτήματα. Κάτι το οποίο ακούσαμε στο τέλος Υπάρχουν ακόμα μέλη του Κοινοβουλίου που θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση μια νέα συνθήκη είναι δυνατή. Εγώ θεωρώ αδύνατο κάτι τέτοιο. Αδιανόητο με πολιτικού όρου θα ήταν να λάβουμε κύρωση από 28 κράτη-μέλη οποιασδήποτε συνθήκη αυτή τη στιγμή, με οποιοδήποτε περιεχόμενο. Σε κάποια κράτη-μέλη χρειαζόμαστε δημοψηφίσματα, όχι στη δική μου, εκεί απαγορεύεται το Σύνταγμα, αλλά χρειαζόμαστε δημοψήφισμα, για παράδειγμα, στη Γαλλία το επίπεδο αποδοχής ε, και δημοτικότητας ε, του Προέδρου Ολάντα αυτή τη στιγμή είναι 13%. Πραγματικά ότι με τέτοια επίπεδα δημοτικότητας ε, μπορεί κάποιος να περάσει μια συνθήκη. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν μπορώ να φανταστώ μια συνθήκη να υιοθετείται με ομοφωνία από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό επικεντρώνομαι όχι μόνο στα μικρά ίσονο σημασία, γιατί υπάρχουν και ουσιώδη πράγματα που μπορούν να γίνουν. Κυρία Μπέσο, ρωτήσατε τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να προσαρμοστεί στη διαφοροποίηση. Ο πρόεδρος Μπαρόσο έκανε μια πρόταση και θα κρυφτώ κι εγώ πίσω από το όνομά του. Για να πω ότι η πρόταση μιας ειδική επιτροπής που θα ασχολείται με ζητήματα του ευρώ είναι μια καλή ιδέα, μπορούμε να εξετάσουμε. Είπατε ότι κάθε κοινοβούλιο εκπροσωπεί και την κοινότητα. Αυτό ισχύει, αλλά πρέπει όλα αυτά να ψηφιστούν στην Ολομέλεια. Μιλάμε, λέμε ότι ε, το βασικό τμήμα των εργασιών του Κοινοβουλίου γίνονται μέσα στις επιτροπές. Νομίζω ότι το Βρετανικό Κοινοβούλιο, που είναι από το παλαιότερα στην Ευρώπη μετά τη Ισλανδίας, έχει μια διαφορετική διαδικασία, γιατί και, τα, ε, και οι Σκοτσέζοι βουλευτές ψηφίζουν επί του αγγλικού, ε, βάσει του αγγλικού δικαίου, ενώ δεν σημαίνει το αντίστροφο με τους ε, Άγγλους βουλευτές και το Σκοτσέζικο δίκαιο. Αυτό είναι όμως ε, ένα ειδικό ζήτημα και μπορούν ε, να βρεθούν και λύσεις. Τώρα, για το σύστημα δύο ταχυτήτων, ξέρω ότι αυτό είναι λεπτό ζήτημα σε πολλά τμήματα της Ευρώπης, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και όχι μόνο πολλών ταχυτήτων και πολλών επιπέδων. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας και στόχων, όπως είναι το ευρώ. Πρέπει να το αποδεχθούμε λοιπόν και να προσαρμοστούμε σε αυτήν την κατάσταση. γιατί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μίλησατε για τους Spitzenkandidat. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό το θέμα θα υπάρξει και στις επόμενες ευρωεκλογέ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εξέτασαν πολύ, τους είναι στη διαδικασία εκλογής των Spitzenkandidaten γιατί είναι κάτι το οποίο θα αξιοποιήσουν στο μέλλον. Τέλος, βεβαίως και είναι τεχνικό το θέμα. Πάντα τεχνικές διαστάσεις υπάρχουν στην πολιτική. Και δεν μιλώ εδώ για, τη βελγική πολιτική σκηνή που έχει πλέον πάρει άλλες διαστάσεις πολυπλοκότητας. Αλλά είναι και αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων να εξηγούν τα πολύπλοκα στοιχεία της πολιτικής με απλό τρόπο. Πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη, μεταξύ των θεσμικών οργάνων, τις σχέσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και τη δυσπιστία που υπάρχει στα κράτη-μέλη για την ε, υπερβολική ε, εξουσία της Επιτροπής. Αυτή είναι η δική τους γνώμη βεβαίως, δεν λέω ότι έχουν δίκιο, αλλά αυτό σκέφτονται. Και υπάρχουν και ζητήματα που πλέον ε, των τεχνικών πτυχών της πολυπλοκότητας υπάρχουν και άλλα πρακτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ε, που απευθύνονται στη κοινή γνώμη, ε, στα θεσμικά όργανα των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου, το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ. Ο καθηγητής Φανσλάμ. Ναι, τέσσερις παρατηρήσεις έχω μόνο, γιατί ακούσαμε πολλά ερωτήματα. Αρχικά, η προβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εθνικό επίπεδο. Εμένα με απασχολεί το ζήτημα της στήριξης. Χάρηκα λοιπόν που τελικά η μέση συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές ήταν πάνω από 40%. Αν ε, είχε πέσει κάτω το 40% θα ήταν πολιτική καταστροφή. Επομένω, αφετηρία μας είναι ο πολίτης που πρέπει να χρησιμοποιήσει, να ε, ασκήσει το δικαίωμα ε, να ψηφίσει σε ευρωπαϊκέ εκλογέ. Έχουμε και εμεί ευθύνη λοιπόν. Τώρα, από εκεί πέρα, η κύρια, την κύρια ευθύνη την έχουν ε, οι πολιτικοί σε εθνικό επίπεδο. Τα μέλη των εθνικών κυβερνήσεων, των εθνικών κοινοβουλίων, θα πρέπει να αναλάβουν ε, περισσότερη δράση ω νέα διάσταση στη διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να εξηγούν τι έχει επιτευχθεί είτε νικούν είτε χάνουν σε ένα τέτοιο πολιτικό διάλογο. Νομίζω όμως ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει περισσότερα, όχι μόνο σε τεχνικά κείμενα, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους νομοθετικές προτάσεις, αλλά και σε δημόσιες ακροάσεις. για να ε, έχουμε και την πλήρη προσοχή ε, των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Είναι δύσκολο, αλλά είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο. Για τον κύριο Λάινεν. Εξαρτάται και από το πώς θα λήξει αυτή η συζήτηση σε ό,τι αφορά ε, τη μορφή της Επιτροπής ως ε, συλλογικό φορέα. Θεωρώ ότι ήταν ιδιοφυής η ιδέα των Spitzenkandidaten θέτει μια νέα διάσταση και στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο, αν αυτές οι ακροάσεις που γίνονται τώρα ε, είναι υπερβολικά πολιτικοποιημένες και δεν επικεντρώνονται τόσο στην ουσία εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσετε τελικά ψήφο εμπιστοσύνη στην Επιτροπή ως σύνολο. Ιδάλλως θα... Ε, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται ακόμα και να επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Για την ενισχυμένη συνεργασία, συμφωνώ με την ιδέα σας ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει τη σταθερότητα και τη συνοχή. Αλλά η ενισχυμένη συνεργασία είναι μια αρχή που ισχύει στο πλαίσιο των στόχων της συνθήκης την οποία έχουν ε, προσχωρήσει όλα τα κράτη-μέλη και αξιοποιείται ως ε, μέτρο τελευταίας ανάγκης, έκτακτης ανάγκης. Δέχεστε, δεχόμαστε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεχόμαστε ότι ε, θα θεσμοθετήσουμε αυτό τον μηχανισμό των δύο ταχυτήτων όπως θέλετε να το πείτε. Προς όφελος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετέχουμε όλοι, πρέπει να εξετάσουμε ακριβώς αυτές τις απαιτήσει και προϋποθέσεις που εγγράφονται και στην ε, συνθήκη του Άμστερνταμ και με την προοπτική της ε, διεύρυνσης με τα 12 νέα μέλη Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και που και πάλι ε, έτυχε καχυποψίας και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, τουλάχιστον στην αρχή, δεν πρόκειται να υπερβούν τις προσδοκίες μας στο μέλλον. Βεβαίως και μπορούν να το κάνουν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερη ευελιξία. Κύριε Άντρεσον, το ίδιο επιχείρημα και στα όσα είπατε εσείς, συμμερίζουμε απόλυτα τη γνώμη σας. Όταν εργαζόμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ακριβώς αυτό υπερασπιστήκαμε και εμείς, ε, την ενότητα, την ομοιομορφία μεταξύ όλων των κρατών μελών. Αλλά όπως ήδη ανέφερα στο ε, Διεθνές Ενωσιακό Δίκαιο, είναι μια παγιωμένη αρχή πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Αυτό είναι προ όφελο των ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα είναι λοιπόν να δώσουμε ένα opt-out σε κάποια κράτη-μέλη, όπω ισχύει και για τη Δανία. Με πλήρε opt-out, το οποίο είναι αποδεκτό αρκεί να επιτρέπεται σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν να το πράττουν. Αυτή είναι η κύρια επίπτωση. Αν έρθουμε αντιμέτωποι και ελπίζω να μην γίνει αυτό, ε, με μία περίπτωση όπου θα ε, αρνηθούμε το δικαίωμα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν επειδή κάποιοι διαφωνούν. Και βεβαίως και είμαι υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι κάθε στιγμή, κάθε Ανά πάσα στιγμή όλα τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να κάνουν τα ίδια βήματα. Γι' αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να το σκεφτούμε. Και ελπίζω να συμφωνήσετε κι εσείς τουλάχιστον να το εξετάσετε, τα υπέρ και τα κατά. Και δέχομαι ότι υπάρχουν και τα αρνητικά. Ευχαριστώ κύριο Σαμανουηλίδης τώρα. Πέντε σημειώσεις. Θα είμαι σύντομος, δεν θα αντιμετωπίσω όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν για τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Όπως ελέγχθη προηγουμένως, έχουμε ήδη μια διαφοροποιημένη Ευρώπη. Και αυτό ήταν θετικό για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, γιατί υπήρξε αυτή η διαφοροποίηση για ένα διάστημα πια. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργηθεί ένα είδος πολλαπλών επιπέδων, μιας ε, αθέλητης διαφοροποίησης μεταξύ πυρήνα και περιφέρειας, όπου ορισμένοι στην περιφέρεια δεν μπορούν να πλησιάσουν την ε, τον πυρήνα. Το να έχουμε μια συνθήκη του ευρώ και μια ένωση του ευρώ, αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω διαιρέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν νομίζω ότι οι χώρε του ευρώ είναι τόσο συνεκτικέ ώστε να μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα μόνο ω χώρε του ευρώ. Δεύτερο, για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αλλά επίση αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχετε ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και δεν μιλάω για τη δημιουργία νέων θεσμών. Αυτό δεν το υποστηρίζω. Απλώ όμω θα πρέπει να βρούμε τρόπου να ενσωματώσουμε τα εθνικά κοινοβούλια περισσότερο στην χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών. Η εφαρμογή συστάσεων αναχώρα βάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αυτό θα είναι κάτι όπου τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ασχολούνται περισσότερο για το θέμα αυτό. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί να κάνει κανείς. Τρίτον, ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι για να βρούμε τι ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε διακρίσεις και αυτό μας ξαναφέρνει στα θέματα της διαφοροποίησης. Θα πρέπει να αποφασίζουμε μονάχα κατά περίπτωση σε σχέση με αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν στο μέλλον, παραγωγικά, υπάρξει δημοσιονομική αρμοδιότητα η οποία εμπλέκει τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη, να υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των βουλευτών που έρχονται από τι χώρε οι οποίε συμμετέχουν σε αυτή τη δημοσιονομική συμφωνία και σε αυτέ που δεν το κάνουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει γενικά, μπορεί να γίνει μονάχα κατά περίπτωση. Τέταρτον ο ρόλο της Γερμανίας. Η Γερμανία παίζει ένα ηγετικό ρόλο, αλλά την έσπρωξαν οι περιστάσει σε αυτόν τον ηγετικό ρόλο. Το 2010 υπήρξαν άλλοι που είπαν στου Γερμανού: Πάρτε ευθύνη, κάντε κάτι, βοηθήστε μας σε σχέση με την κρίση αυτή, η οποία γίνεται όλο και χειρότερη. Οι Γερμανοί στην αρχή ήταν διστακτικοί, δεν θέλανε να αναλάβουν αυτό τον ρόλο, κάποια στιγμή τον ανέλαβαν. Και είπαν όλοι, μα δεν θέλαμε να το κάνετε αυτό. Αλλά έτσι γίνεται μερικέ φορέ. Έχουμε τώρα μια κατάσταση όπου οι Γερμανοί ασκούν αυτόν τον ηγετικό ρόλο, αλλά είναι πολύ δύσκολο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για του ίδιου του Γερμανού. Μερικέ φορέ θα πρέπει να βρούμε τρόπου να βοηθήσουμε του Γερμανού σε αυτόν το ρόλο ηγεσία, δηλαδή να τον εξισορροπήσουμε καλύτερα με το να ενισχύσουμε άλλα κράτη-μέλη όπω είναι παραδείγματο χάρη η Γαλλία, να βρούμε άλλε συμβαστικέ λέσει. Και αυτό που είπε ο Φιλίπ και αυτό που είπε ο κ. για ένα φαινόμενο που κάποιος ονόμασε έλλειψη εμπιστοσύνης και κάποιος άλλος ονόμασε ανισότητες. Εγώ μίλησα για θρημάτιση, για κατακαιρμάτιση, αλλά είναι περίπου το ίδιο θέμα. Το ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη, την κατα... κατακαιρματισμό, την ε, έλλειψη εμπιστοσύνη είναι κατακαιρματισμό σε οικονομικό, σε πολιτικό, σε κοινωνικό επίπεδο μέσα στα κράτη-μέλη και μεταξύ των κρατών μελών. Πώ θα το αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτό, και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ περισσότερο γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει πανάκια. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτό που είπαμε προηγουμένω, μια συνολική συμφωνία, ένα new deal, μια νέα συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών που προσπαθεί να εξορροπήσει τα συμφέροντα των κρατών μελών. Δηλαδή πρέπει να εντοπίσουμε αυτά τα οποία είναι σημαντικά και για τι 28 χώρε και να δημιουργήσουμε μια συνολική λύση. Η συνολική λύση δεν είναι αλλαγή των συνδικών, μπορεί να είναι μια πολιτική συμφωνία θα πρέπει να βρούμε όμως τα στοιχεία αυτά τα οποία θα καλύψουν τα διαφορετικά, τα αποκλίνοντα εθνικά συμφέροντα. Εγώ δεν παρακολούθησα αυτά που είπε ο κύριος Κατάναν για, το, για την χάτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά αν ακολουθήσει κανείς τέτοιο δρόμο κάνει λάθος. Ένα στοιχείο αυτής της νέας συμφωνίας θα πρέπει να είναι να βοηθήσετε την αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την φροντίδα και προστασία ότι υπάρχει μια κοινωνική βάση η οποία πάντα θα διατηρηθεί. Αν πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση στις χώρες σε οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει ένα ελάχιστο το οποίο θα διατηρηθεί και το οποίο θα μειώσει το φόβο ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι ένας αγώνας ανταγωνισμός προς το χειρότερο. Νομίζω λοιπόν ότι ένα τέτοιο σύμφωνο για να έχει νόημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα νέο όραμα, ένα νέο εγχείρημα, κάτι το οποίο λειτουργήσε πολύ καλά στο παρελθόν όταν είχαμε αδιέξοδο. Δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκεται αυτό, μπορεί να είναι η ενέργεια ή κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Ε, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε. 6 ε, Νοεμβρίου η επόμενη συνεδρίασή μας αγαπητοί συνάδελφοι και έχουμε ε, την ακρόαση αύριο. Ελπίζω ότι θα είστε όλοι παρόντες. Ευχαριστώ.